So, colleagues, I think we can start, despite the empty room. Not, not completely empty, but still. Uh, hopefully our colleagues will come later, but let's time to... Uh... Καλημέρα σας, ας αρχίσουμε. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης, στάλη. Υπάρχουν αντιρρήσεις, αν όχι, μπορεί να εγκριθεί. Δεύτερο σημείο, έγκριση των πρακτικών από 20-21 Ιανουαρίου. Έχει, έχουν σταλεί στα μέλη της Επιτροπής. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορούν και αυτά να εγκριθούν. Ωραία. Ευχαριστώ. Σημείο 3. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Δεν έχω να πω τίποτε, εκτός από το να καλημερίσω όλους σας. Σημείο 4 μια έκθεση της ΕΟΚΕ για τα δικαιώματα τα εκλογικά των ανθρώπων με αμα αναπηρία. Εκατομμύρια άνθρωποι δεν επιτρέπεται, δεν μπορούν να ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Εδώ έχουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Πάτερ. Θα σας δώσω το λόγο για 10 λεπτά και μετά την παρουσίαση θα κάνουμε ερωτήσεις για 15 λεπτά περίπου. Εγώ είμαι από την Εστονία. Ξέρω δηλαδή ότι ένα λεπτό είναι 60 δεύτερα. 10 και 15 λεπτά λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ που με καλέσατε και μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτή την έκθεση για τα πραγματικά δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες να ψηφίζουν. Από το Μάρτιο του 19 είναι η έκθεση. Δείχνει ότι έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη. Θα σας εξηγήσω. Η έκθεση είναι μια ιστορία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζει το πραγματικό της πρόσωπο και δυστυχώς το πρόσωπο αυτό δεν είναι φωτεινό. Ε, δείχνει ότι εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρία δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές. Ποιος ήταν ο στόχος της έκθεσης. Ο στόχος ήταν να παρουσιάσουμε την πραγματική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, ευρωεκλογές. Η Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΟΚΕ μπορεί να αποφαίνεται για θέματα που αφορούν την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Περίπου δύο χρόνια χρειάστηκε η έκθεση. Η διαδικασία συλλογής δεδομένων ήταν περίπλοκη. Εγώ ήθελα να δείξω την κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης με την εξαίρεση του Ηνωμένου Βασιλείου γιατί εκείνη την εποχή ήταν, ε, θεωρούσαμε ότι δεν θα συμμετείχαν στις εκλογές. Η διαδικασία συλλογής ε, αποτελείται από δύο έρευνες. Η μία συλλογή δεδομένων σε σχέση με τους περιορισμούς, δηλαδή ε, φραγμή και τεχνική φραγμή. Οι περισσότερες απαντήσεις που ελάβαμε ήταν από δημόσιες αρχές ή οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών που εστιάζουν στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα ανθρώπων με αναπηρία. Υπάρχουν πάνω από 200 παραδείγματα από όλα τα κράτη-μέλη. Τα θετικά παραδείγματα παρουσιάζονται μαζί με το όνομα του κράτους μέλους, ενώ τα αρνητικά παραδείγματα παρουσιάζονται ανώνυμα, γιατί η έκθεση δεν, είναι να δεν έχει σκοπό να επικρίνει, απλώς να καταδείξει τα προβλήματα. Το σημείο αφετηρίας της έκθεσης είναι να αναφερθεί στα βασικά διεθνή νομικά και πολιτικά ε, πλαίσια, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Προσώπων με Αναπηρίες, ε, ε, έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Επίσης παρουσιάζεται και το ιστορικό πλαίσιο όπως και λεπτομερείς κανόνες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκλογές. Και βλέπουμε πώς μπορούν να εξελιχθούν αυτοί οι κανόνες για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα άτομα με αναπηρία. Καταρχήν η νομική φραγμή στέρηση εκλογικών δικαιωμάτων πριν από 20 χρόνια υπήρχε μια κοινή θέση ότι άνθρωποι με ψυχικά προβλήματα ε, δεν είχαν ε, την νομική ικανότητα να συμμετέχουν στις εκλογές. Τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σε 12 συν 2, δηλαδή τελευταία στιγμής αλλαγές που έγιναν στις αρχές του 2019 στη Γερμανία και τη Γαλλία αυτό αυτόματη απώλεια δικαιωμάτων ε, ψήφου ε, όταν δεν υπάρχει νομική ικανότητα 9 1 και αξιολόγηση που γίνεται με βάση την ικανότητα του ατόμου 7 1, δηλαδή 6 κράτη-μέλη κάνουν αξιολόγηση αλλά λάβετε υπόψη ότι σε αυτή την ομάδα υπάρχει μια χώρα Ε, που έχει μόνο 100 περιστατικά, ενώ μια άλλη έχει 40.000 ε, περιστατικά. Ε, τεχνική φραγμή σε 8 κράτη-μέλη, πληροφορία για την εκλογική διαδικασία είναι πολύ περιορισμένη και παρέχεται μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου. Δεν υπάρχει προσαρμογή στις ανάγκες ανθρώπων με συγκεκριμένες αναπηρίες. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκλογικών τμήματων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν προσαρμοστεί πλήρω ή γενικώ προ τι ανάγκε ανθρώπων με διάφορα είδη αναπηριών. Και σε 12 κράτη-μέλη τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να αλλάξουν εκλογικό τμήμα αν σε ένα άλλο εκλογικό τμήμα είναι καλύτερα τα πράγματα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Κανένα κράτος μέλος δεν έχει τυποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο τα εκλογικά τμήματα είναι εξοπλισμένα και λειτουργούν για να είναι φιλικά προς τον χρήστη για όλους τους εκλογείς. 50% ε, ή στο, στο Βέλγιο ε, υπάρχουν κάποιες οδηγίες που δημοσιεύονται από τις τοπικές αρχές ελεύθερη επιλογή ενός βοηθού δεν επιτρέπεται σε κάποια κράτη-μέλη. Μόνο σε εννέα κράτη-μέλη οι τυφλοί μπορεί να ψηφίσουν με πλήρη μυστικότητα και χωρίς καμία βοήθεια. Σε όλα τα άλλα δεν επιτρέπεται. Είναι αδύνατον σε κάποια κράτη-μέλη η διαδικασία της ΦΥΦΟΥ. Δεν είναι εύκολο να γίνει κατανοητή από τους εκλογείς, οπότε δεν καταλαβαίνουν τις συνέπειες συγκεκριμένων μεθοδολογιών ψήφου και καλούνται να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα για να ψηφίσουν, όπως να γράψουν το πλήρες όνομα του υποψηφίου που θέλουν να ψηφίσουν. Στο 1 τρίτο περίπου των κρατών μελών, οι άνθρωποι που διαμένουν συνεχώς σε ιδρύματα ή σε νοσοκομεία δεν έχουν δυνατότητα να συμμετέχουν στις εκλογές. Τώρα κάποια άλλα θέματα που παρουσιάζονται στην έκθεση που δεν θα αναφέρω λεπτομερώς αλλά υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας και στα έγγραφα που αφορούν τη σημερινή έκθεση. Συζητήθηκε η ψήφος νωρίς, ταχυδρομική ψήφος, ψήφος με κινητή κάλπη, ε, διαντιπροσώπου, δεν νομίζω ότι είναι εναλλακτική η ψήφος δια ε, αντιπροσώπου, γιατί είναι μεταβίβαση εκλογικού δικαιώματος. Μπορεί να είναι συμπληρωματική μονολύση. Η ηλεκτρονική ψήφος υπάρχει, προβλέπεται δηλαδή σε δύο κράτη-μέλη στο ένα αποπλήρωσε, σε ένα άλλο όχι απόλυτα, αλλά πάντως υφίσταται. Υποχρεωτική ψηφοφορία σε, τρεις, σε τρία κράτη-μέλη. Είναι υποχρεωτική συμμετοχή στις εκλογές, εκτός και αν ε, δεν έχουν τη δυνατότητα. Κάποια βασικά συμπεράσματα. Σε κάθε ένα από τα 27 κράτη-μέλη υπάρχουν νόμοι ή οργανωτικές ρυθμίσεις που αποκλείουν ορισμένους ψηφοφόρους με αναπηρίες από τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές περίπου 400.000 πολίτες της Ένωσης από 14 κράτη-μέλη ε, λόγω εθνικών κανόνων στερούνται το δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωεκλογές λόγω της αναπηρίας τους ή των ψυχικών προβλημάτων, ψυχικών προβλημάτων ψυχικής υγείας. 800.000 ήταν αυτοί πλέον τις αρχές του 2019. Αλλά επειδή κάποια κράτη-μέλη εξαιρούνται, πήγαμε στι 400.000. Σε 8 κράτη-μέλη κάποιο που δεν μπορεί να πάει σε εκλογικό τμήμα δεν μπορεί να ψηφίσει γιατί δεν έχει την εναλλακτική ε, δυνατότητα ψήφου. Όπω είπα, σε 18 κράτη-μέλη οι τυφλοί ψηφοφόροι δεν μπορούν να ψηφίσουν ανεξάρτητα, αυτόνομα. Αν οι βέλτιστες πρακτικές από όλες τις χώρες εφαρμόζονταν, θα δημιουργούνταν ένα ιδανικό σύστημα όπου κάθε πολίτης της Ένωσης με αναπηρίες όχι μόνο θα είχε 100% δυνατότητα ψήφου, αλλά θα μπορούσε να επιλέξει τον πιο ε, βολικό τρόπο για να ψηφίσει. Η τρέχουσα ε, νοσιακή νομοθεσία ήδη ασχολείται με έναν αριθμό θεμάτων που αφορούν τις ευρωεκλογέ. Έτσι δεν υπάρχουν τυπικά εμπόδια στην νομοθεσία αυτή, συμπεριλαμβάνοντας και εγγύησεις για τις εναλλακτικέ επιλογές ε, για την ψηφοφορία ατόμων με αναπηρία. Θα πρέπει να είναι διασφαλισμένο το δικαίωμα ε, συμμετοχής στις εκλογές για ανθρώπους με ψηφοφορία. Ε, αυτή τη φορά ψηφίζω. Ε, αυτό ήταν το σλόγγαν για τις τωρινές ευρωεξο, Αλλά δυστυχώς πολλοί άνθρωποι με αναπηρία ε, θα έλεγαν αυτή τη φορά πάλι δεν μου επιτρέπεται να ψηφίσω. αυτή η έκθεση αφορά τον γκρίζο πρόσωπο της Ένωσης, Όμω το μέλλον μπορεί να είναι φωτεινό για όλους. Τώρα είναι ώρα για δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δέχτηκε το αίτημά μου να εργαστώ πάνω σε μια έκθεση πρωτοβουλίας για αυτό το θέμα. Και θέλω να καταδείξω σε μια πολύ σύντομη γνωμοδότηση τι πρέπει να αλλάξει στον εκλογικό κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλιστεί ότι η πλειοψηφία τουλάχιστον των ανθρώπων με αναπηρία θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εκλογές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ εντυπωσιακά και πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Θα δώσω πρώτα τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και φοβάμαι ότι δεν θα πω το όνομά σας ε, σωστά. Πάντως, σας δίνω τον λόγο. Δεν πειράζει. Η Μακουλάδα Πλαθένθια Πορέιρο λέγομαι και εργάζομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην ε, μονάδα που ασχολείται με την ε, απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Πάθρα γιατί πρόκειται εδώ για μια εξαιρετική γνωμοδότηση που περιλαμβάνει πάρα πολύ σημαντικά ε, πληροφοριακά στοιχεία και που ανταποκρίνεται ή συστοιχίζεται πολύ σωστά με τις πληροφορίες τις οποίες έχει συλλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είτε με την υπηρεσία ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων είτε μέσω εξωτερικών συνεργασιών. Και εδώ μιλάμε βέβαια για τις δυσκολίες σχετικά με την ψήφο Ωστόσο δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία υπογραμμίζει το γεγονός της πολιτικής συμμετοχή σε οποιοδήποτε επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβληματιστεί ε, για το θέμα αυτό μετά από το ξεκίνημα της στρατηγικής ε, για τα άτομα με αναπηρία. Έχουμε λάβει ε, υπόψη μας τα στοιχεία αυτά, αλλά ε, μαζί με τους εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες ε, των κρατών μελών ε, στην ομάδα υψηλού επίπεδου για την αναπηρία. Και κατά την έννοια αυτή θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι, ο, ε, ότι η οδηγία και η πράξη ε, για την προσβασιμότητα θα βελτιώσουν πάρα πολύ την κατάσταση ε, καθώς επίσης και τα θέματα τα οποία αφορούν την τυποποίηση για το οικοδομημένο περιβάλλον. Επίσης ε, και ε, στην ε, περίπτωση των ευρωπαϊκών εκλογών είχαμε σημειώσει τα τα ενδεχόμενα προβλήματα σε σχέση με τη δυνατότητα ψηφοφορίας. Αυτή τη στιγμή ε, αξιολογούμε την, ε, στρατηγική, ε, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αναπηρία και τα άτομα με αναπηρία και οπωσδήποτε αυτό θα αποτελέσει και τροφή για σκέψη και στο μέλλον, για το μέλλον της στρατηγικής αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Ανταμ Κόζατς. Δεν ξέρω αν έχει ερώτηση προς την Κομισιόν, προς τον εισηγητή, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε κύριε Πάτερ σε αυτήν την ε, συνεδρίαση. Εμεί ε, βεβαίως είμαστε από καιρό σε επαφή, έχετε έρθει επανειλημμένα, έχουμε βρεθεί και ε, βεβαίως συζητούμε και με διάφορες ε, επιτροπές, με διάφορους ε, με διάφορες οργανώσεις για την ουσία του θέματος. Το έγγραφό σας το διάβασα και καταλαβαίνω ότι αντιμετωπίζουμε δύο προκλήσεις, μία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μία σε επίπεδο κρατών μελών, σε σχέση με το ενωσιακό επίπεδο σε αυτήν την έκθεση εδώ μιλάμε για τις ευρωπαϊκές εκλογές και η πρόκληση είναι η εξής. Σε όλα τα κράτη-μέλη μπορούμε να καταφέρουμε ε, η ψηφοφορία να γίνει χωρίς ε, ε, κανένα εμπόδιο. μέσα από ε, μεταρρύθμιση των θεσμών. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ε, και τεχνικά προσκόμματα. Ξέρετε ότι υπάρχουν κανόνες που σχετίζονται με, την, με τις εκλογές ε, και που αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Άρα είναι δύσκολο να προκύψει εναρμόνιση όσον αφορά αυτούς τους κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν το, ε, το Κοινοβούλιο μέσω της εκθέσεώς του να καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει αποφασιστικά μέτρα έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να αρχίσουν διαπραγματεύσεις όσον αφορά αυτά τα ζητήματα έτσι ώστε να προκύψουν εναρμονισμένες κατελάχιστον τουλάχιστον ε, κανόνες δηλαδή να υπάρξουν ελάχιστες εγγυήσεις ε, σε όλες τις χώρες έτσι ώστε άνθρωποι με αναπηρία να μπορέσουν να πάνε να ψηφίσουν ψηφίσουν χωρίς προσκόμματα. Ευχαριστώ. Maybe, ίσως να απαντάτε σε κάθε μία ερώτηση. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα βρίσκεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράδειγμα, Ευρωπαϊ... Ευρωπαίος πολίτης με δύο διαβατήρια έχει δικαίωμα, μπορεί να έχει ή να μην έχει δικαίωμα να ψηφίσει στις ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτό που περιμένουμε εμείς σαν ΕΟΚΕ και το έχουμε εκφράσει είναι να υπάρξει διασφάλιση βασικών δικαιωμάτων και ε, εγγυήσει να παρέχονται για τα βασικά δικαιώματα σε, όλα τα, σε όλους τους πολίτες. Ε, γιατί αν πούμε, ας πούμε, ότι κάθε τυφλός θα πρέπει να ε, διασφαλίζει το δικαίωμά του να ψηφίσει ε, ε, χωρίς πρόβλημα και μυστικά, τότε Ε, θα πρέπει για τις ευρωπαϊκές εκλογές να τροποποιηθεί το σύστημα ε, ε, κατά αναλογικότητα. Έχει λοιπόν την δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει τους κανόνες. Τέλος. Στην περίπτωση της Δανίας να αναφερθώ. Η Δανία βάσει συντάγματος έχει διάταξη που δεν επιτρέπει ε, σε άτομα τα οποία δεν έχουν, ε, ε, πολιτικά, δεν έχουν τα πολιτικά τους δικαιώματα να ψηφίσουν για τις ευρωπαϊκές εκλογές και για τις τοπικές εκλογές. Ορισμένες όμως χώρες έχουν ε, περιορισμούς λοιπόν. Ερώτηση, αυτή, αυτός ο περιορισμός εφαρμόζεται πάντα για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Έχω, ε, διατηρώ επιφυλάξεις και αμφισβητήσεις. Απ' την άλλη πλευρά, οι τεχνικές, ε, τα τεχνικά εμπόδια μπορούν να έρθουν αρκετά εύκολα. Ευχαριστώ. Προσωπικά, προσωπικά πιστεύω ότι η πρόταση είναι πολύ και είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε στην Επιτροπή μας και ως Επιτροπή Αναφερών να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο θέμα. Κύριε Σορόρα. Κύριε, κύριε Ο κύριος Μάριο Φουρόρα, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον αυτήν ε, την ε, έκθεση. Ε, κοινωνικές μάχες έχουν δοθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο το δικαίωμα ψήφου. Πρόκειται για ένα δικαίωμα το οποίο αναγνωρίζεται σε όλους ε, χωρίς καμία διάκριση βασισμένη στο φύλλο, τη θρησκεία ε, ε, ή οτιδήποτε άλλο. Όμως 800.000 και πλέον πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα κράτη-μέλη ε, της ε, Ιδίας δεν έχουν την δυνατότητα να ψηφίσουν. Ε, απ' την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι διαπιστώνουμε μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις συμβάσεις οι οποίες δεν εφαρμόζονται σωστά. Στην χώρα μου την Ιταλία αναγνωρίζεται το πλήρες δικαίωμα στην ψήφο και επομένως επομένως ελπίζουμε ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται και να επιτρέπεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά δια αντιπροσώπου ε, ε, με επιστολική ψήφο κλπ. Ακόμα και μέσα ε, στα νοσοκομεία. Εγώ προσυπογράφω τα όσα είπε ο προλεγγύης συνάδελφος και νομίζω ότι είναι απαραίτητο τουλάχιστον το 2024 όταν θα γίνουν οι επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές όλοι να έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν σύμφωνα με τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο. Στο παιχνίδι αυτό, αν θέλετε, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο τρόπος είναι πολύ απλός. Οι αλλαγέ στον εκλογικό κώδικα για τι ευρωεκλογέ εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά εγκρίνονται στο επίπεδο του Συμβουλίου από τα κράτη-μέλη. Και λύθηκε το πρόβλημα. Το πρώτο σκέλος λοιπόν είναι, το πρώτο στάδιο. Αυτή τη στιγμή συγκριθεί η έκθεση από την ε, ΕΟΚΕ, αυτή να αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έγινε αυτό, το θέμα είναι πώς θα δώσουμε εμείς συνέχεια. Υπάρχουν ερωτήσεις από τους συναδέλφους, αλλά έχω και εγώ μία. Αντιλαμβάνομαι ότι μιλούμε για άτομα με αναπηρία, αλλά επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχουν και πολίτες μεγάλης ηλικίας οι οποίοι μπορεί να μην έχουν αυτό το στάτους επίσημα, αλλά έχουν κάποιες δυσκολίες, αν όχι αντίστοιχες με το άτομα με αναπηρία. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για αυτούς. Δεύτερον, αναφέρατε ότι υπάρχουν δύο κράτη-μέλη στα οποία υφίσταται ηλεκτρονική ψήφο και είπατε για την ακρίβεια ότι ένα από τα δύο μπορεί να γίνει ε, ψήφο μέσω ίντερνετ. Πόσο ακριβώ λειτουργεί αυτό, Μιλάτε για την Εστονία, για την ηλεκτρονική ψήφο που έχουμε στην Εστονία και πόσο αυτό βοηθά τα άτομα με αναπηρία. Δεν, δεν το γνωρίζω, θα θέλω να μου το εξηγήσετε. Πρώτα απ' όλα για μένα, άτομα με αναπηρία είναι όλα εκείνα που θα πρέπει να τύχουν της προστασίας που τους δίνει η σύμβαση των ατόμων με αναπηρία, το οποίο, δεν σημαίνει, το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει μια ιδιαίτερη απόφαση αναγνώρισης του ειδικού νομικού στάτους. Συμπεριλαμβάνεται λοιπόν και οι πολίτες μεγάλης ηλικία δικαιωμένοι. Ε, συμπεριλαμβάνονται για παράδειγμα άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους ή επειδή βρίσκονται σε κάποιο ε, ε, θεραπευτήριο. Αυτοί δεν μπορούν να συμμετέχουν στις ευρωεκλογέ. Στην Εστονία λοιπόν τώρα για την ηλεκτρονική ψήφο ε, υπάρχουν κάποια μηχανήματα εγκατεστημένα μόνο σε ορισμένα εκλογικά τμήματα. η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων μεταξύ του πολίτη και του κράτους είναι ένα πολύ διαδεδομένο, μια πολύ διαδεδομένη κατάσταση στην Εστονία. Δεν είναι κάτι που χρησιμοποιούμε μόνο για τις εκλογές. Επομένως είναι γνωστό στους πολίτες. Και έτσι, εάν βρεθούν σε μια κατάσταση που δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους, δεν μπορούν να μετακινηθούν, χρησιμοποιούν αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα για να επικοινωνήσουν με το κράτος, για το, με τη δημόσια διοίκηση. Και ορισμένοι από αυτούς το χρησιμοποιούν και για τις εκλογές. Όμως, εγώ σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι η ηλεκτρονική ψήφο, τα ηλεκτρονικά συστήματα μπορούμε να τα θεωρήσουμε μοναδική και πλήρη λύση. Όπως έλεγα, για πολλούς ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό για την ιδιότητά τους ως πολίτες να, να, να αισθάνονται ότι μπορούν να πάνε στο εκλογικό τμήμα και να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Το θεωρούν ε, ύψιστο καθήκον και δικαίωμα. Ε, οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο εκλογικό τμήμα θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες συνθήκες σε αυτό το εκλογικό τμήμα έτσι ώστε να μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους χωρίς να χρειάζεται βοήθεια από κάποιο τρίτο. Ε, ε, εκτός εάν εκείνοι το επιθυμούν βεβαίως. Αλλά ε, το σημείο εκκίνησής μας θα πρέπει να είναι αυτό ως, ως βασική αρχή. Γιατί για, για εμένα είναι ζήτημα ανθρώπινας αξιοπρέπειας, πολύ σημαντική. Χρειάζονται όμως ψηφιακές δεξιότητες. Αν είναι κανείς 82 ετών, δεν είναι τόσο καλός σε αυτές τις δεξιότητες. Η κυρία Στανόκα, ορίστε. Θέλω να πω μόνο ότι καμιά φορά ζητάμε από άλλα κράτη-μέλη περισσότερα από ό,τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Εγώ ήμουν παρατηρήτρια σε πολλές εκλογές ως μέλος της αποστολής παρακολούθησης των εκλογών. συμπληρώνεται ας πούμε η προσπελασιμότητα των εκλογικών τμήματων σε αυτά που παρακολουθούμε που αποτρέπει τους ανθρώπους με αναπηρία. Συχνά ασκείται κριτική για τη μη πρόσβαση. Αυτό το είχα δει στις χώρες ε, του ΟΑΣΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται αυτό. Εμείς παίρνουμε πληροφορίες από δημόσιες αρχές πριν από τις ευρωεκλογέ. Κυρίως για τα εκλογικά τμήματα. Οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνε για την προετοιμασία των εκλογικών τμήματων και πολύ συχνά δεν τα προσαρμόζουν στις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία αλλά ειλικρινά δεν ξέρουν και τι να κάνουν. Ακόμα και αν κάποιος ξέρει τι πρέπει να γίνει, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί καμιά φορά χρειάζονται ε, περισσότερες δαπάνες που δεν τις κάνουν. Τα βασικά πρότυπα σε εθνικό επίπεδο πρέπει να εφαρμόζονται σταδιακά. Στη χώρα μου αυτό ισχύει για το 50% των εκλογικών τμήματων. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει δικαίωμα, αν ε, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τα πράγματα κατά 100%. Μπορούμε να πάμε σιγά σιγά, να εξασφαλίσουμε τη μεταφορά τους εκεί. Αλλά δεν κάνουν πολλές φορές ένα μικρό βήμα ε, για να ξεπεράσουν εμπόδια όπως σκάλες κλπ. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Σίγουρα θα συνεχιστεί και η συζήτηση. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Κομισιόν που έχει δύσκολο όνομα και δεν μπορώ να το πω. Ευχαριστώ και όσους συμμετείχαν στη συζήτηση. Πάμε τώρα στην ψηφοφορία. Αν συμφωνείτε, Προτιμώ να ψηφίσουμε με τις ηλεκτρονικές μας κάρτες. Πρώτη φορά προεδρεύω ε, σε ψηφοφορία. Ε, δεν ξέρω αν θα μπορώ να ελέγχω τα υπέρ και τα κατά κάθε φορά, οπότε ας αρχίσουμε ηλεκτρονικά από την αρχή. Να κάνουμε έναν έλεγχο πρώτα. Υπάρχει μια πρόταση από τη Γραμματεία να κάνουμε πρώτα έναν έλεγχο για να δούμε αν λειτουργούν όλες οι κάρτες. Ποιο, ποιος είναι ο πιο όμορφος ε, ε, εδώ στην αίθουσα. αρχίζουμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Λειτουργούν όλα. Ψηφίζομαι γνωμοδότη σχετικά με την παρακολούθηση εφαρμογής του νόμου του 2017 και του 2018 της Ένωσης σχέδιο νομοδότησης ε, Ο κύριος Ρουίς Ντεβέσα είναι ο εισηγητής, δεν είναι εδώ, δεν θα μιλήσει λοιπόν. Προχωρούμε, ψηφίζουμε. Συμβιβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική 2. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Συμβιβαστική τρία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16 σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μέρος 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μέρος 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται επίσης. Τροπολογία 18. Αρχίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μέρος 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 47 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 48 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 52. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 56. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τέλος, το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφοι. Τώρα αν κάποιος θέλει να φύγει από την αίθουσα, ας το κάνει τώρα. Και εμείς θα προχωρήσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Όχι, δεν είναι το 5, συγγνώμη. Το σημείο 6 είναι τώρα. So, colleagues, I'm trying to give... Συνάδελφοι, προσπαθώ τώρα να ε, δώσω τον λόγο στον εαυτό μου, αλλά δεν θέλω και να ξυλαριάζομαι, οπότε παρακαλώ, ηρεμήστε. Καθίστε. Please do so. So the next point of the agenda is the opinion to the own initiative report on the situation of fundamental rights. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την κατάσταση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα 18-19. Είμαι η συγκήτρια, γνωμοδότηση εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών. Γι' αυτό θα σας τα πω εγώ ίδια. Δεν είχαμε πολύ χρόνο και η γνωμοδότηση είναι και πολύ σύντομο κείμενο. Ε, κρίμα για τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, πιστεύω ότι μέσω των τροπολογιών μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Υπάρχουν έξι τροπολογίες. main points. Έξι μάλλον κεντρικά σημεία τα οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω. Ένα είναι το γεγονός ότι η χρήση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, από τις χώρες, ας το πούμε απλά, δεν δεν είναι τέλεια. Ε, επίσης, σημειώνουμε ανησυχία ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν εφάρμοσαν πλήρω ή δεν εφάρμοσαν σωστά την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2008 για την καταπολέμηση ορισμένων ομορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβία μέσω του ποινικού δικαίου. Τρίτον, Θέλω να τονίσω ότι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η ελευθερία έκφραση και ενημέρωση και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωση αποτελούν βασικέ συνιστώσει του κράτου δικαίου και εδώ έχουμε κάποια προβλήματα σε ορισμένε χώρε μέλη. Επίσης, καλούμε την Επιτροπή να εφαρμόσουν τις αρχές του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, έτσι ώστε να κατοχυρωθούν τα κοινωνικά θεμελιώδη δικαιώματα σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, επισημαίνουμε ότι απαιτούνται περαιτέρω διασφαλίσει για την κατοχύρωση και προστασία ιδιωτικής ζωής και τέλος, και αυτό είναι το έκτο σημείο της γνωμοδότησης, καλούμε το Συμβούλιο να ολοκληρώσει με διαδικασία κατεπίδοντας την κύρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Κωνσταντινούπολη Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ε, και εκφράζει την ανησυχία ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν έχουν εφαρμόσει σωστά ή έχουν εφαρμόσει μόνο εν μέρη τη σύμβαση αυτή. Επομένως, ε, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει την νομοθεσία εφαρμογής. Αυτά είναι τα στοιχεία. Ωστόσο, πιστεύω ότι με την βοήθεια των πολιτικών ομάδων και των σκιωδών εισηγητών, θα καταφέρουμε ε, να ε, βελτιώσουμε και σε εύρος και σε βάθος την γνωμοδότηση. Θα δώσω το λόγο στους Κιώδης. Ο κύριος Λοράνι Σέπτο Έλκ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω ουγγρικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρία Τόμα για την εργασία που κάνετε όσον αφορά αυτή την γνωμοδότηση. Εδώ γίνεται λόγος για πολύ σημαντικά πράγματα το είπατε κι εσείς η ίδια ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, γνωμοδότηση και μέσω προτάσεων τροπολογιών. Άλλωστε αυτή είναι η συνήθις διαδικασία του Κοινοβουλίου. Εξετάζουμε την γενική κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέποντας την έκθεση προηγουμένων ετών διαπιστώνουμε ότι πολλά πράγματα δεν έχουν αλλάξει και υπάρχουν ομάδες εντός, της, ε, εντός του κοινωνικού συνόλου που δεν καταφέρνουν ε, να ε, χαίρουν ε, πλήρως των θεμελιδών τους δικαιωμάτων. Υπάρχουν ε, μελέτες ε, και στοιχεία για τα κρατημέλη ε, και οπωσδήποτε τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι. Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και από τον υψηλό ρυθμό αναφορών που φτάνουν στην Επιτροπή μας και είναι σαφές ότι υπάρχουν ακόμα πολλά ζητήματα ε, στη διάρκεια των ε, τελευταίων ε, χρόνων και αποδεικνύεται και από την έκθεση υπάρχουν προβλήματα τα οποία αφορούν την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ρατσισμός, ξενοφοβία, φιλετικό μίσος με διάφορες μορφές ε, ναι, είναι γεγονός, μπορούμε να το πούμε πλέον, υπάρχει ρατσισμό σε πολλές χώρες ε, και μπορούμε να διαπιστώσουμε μάλιστα ότι υπάρχει μια σχετική τάση σε πολλές χώρες. Θα υπάρξουν τροπολογίες γι' αυτό. Επίσης, παραβιάσεις όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το αναφέραμε προηγουμένως σε σχέση με τα εκλογικά τους δικαιώματα, αλλά υπάρχουν προβλήματα και όσον αφορά τα κοινωνικά τους και άλλα δικαιώματα. Πρέπει οπωσδήποτε να τα σημειώνουμε αυτά. Πιστεύω ότι μεταξύ των διαφόρων ε, θεμάτων προκύπτουν διάφορα ερωτήματα τα οποία συνδέονται με τις μειονοτικές ομάδες στην Επιτροπή μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πρέπει να συζητούμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα, πρέπει να προσπαθούμε ε, για την καλύτερη εφαρμογή τους, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας ε, σε αυτήν την διαδικασία. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Γενικά χρειαζόμαστε μια ευνοϊκότερη στάση των κρατών έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα τα οποία επιμένουν και εξακολουθούν να υφίστανται. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα την ευηκονούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα διαβάσει και θα καταλάβει όλα τα στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε τούτη την γνωμοδότηση και που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων, γιατί η η η διασφάλιση των ε, δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ ε, σημαντική και ευελπιστούμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέντσα. Η Κριστίνα μας ε, δεν είναι εδώ από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, επομένως θα δώσω τον λόγο στην Τατιάνα Σντάνοκα που είναι εκπρόσωπος των Πρασίνων εδώ, συντονιστή Σκιώδης. Υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αναφέρεται και στην πρώτη παράγραφο του προσχεδίου γνωμοδότησης αυτό. Και ιδιαίτερη σημασία έχει το άρθρο 51 του χάρτη. που περιγράφει και τις συνθήκες επί τις οποίες μπορούν να περιοριστεί η εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και γνωρίζουμε ότι αυτές είναι σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ ευρείες. Έχει εξάλλου εγκρίνει και ψηφίσματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας τροποποίηση του άρθρου 51 κάτι που θα έδινε περισσότερες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάζει κατά πόσον τα κράτη-μέλη της εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Το είχαμε αναφέρει αυτό και στο ψήφισμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εισηγητή τον κύριο Φερχόφστατ. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν σκόπιμο να το αναφέρουμε και εδώ αυτό το πρόβλημα. Συμμερίζουμε επίσης την ανησυχία που εκφράζει το κείμενο αυτό για το γεγονός ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά επίσης θα ήθελα να υπάρχει και κριτική έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να ζητούμε δηλαδή η Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί περισσότερο και να εκφράζει δημόσια την, ε, ε σε επικρίσεις της για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. να μην επικαλείται τόσο συχνά το άρθρο 51 στις απαντήσεις της προς εμάς ε, και την Επιτροπή μας, ισχυριζόμενοι ότι όλα αυτά δεν είναι αρμοδιότητα της Ένωσης. Είναι ήδη πολύ καλό το κείμενο και ελπίζω ότι θα το βελτιώσουμε την περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Στάνοκα. Από το ECR, ο κύριος Τζαμπάνσκι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε για το προσχέδιο της γνωμοδότησης που μας υποβάλλεται. Έχει καλύψει πολλά σημαντικά θέματα, όμως εγώ αντιπίζω και κάποιες αντιφάσεις. Ιδίω, όταν ζητείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, υποβάλει, να επιβάλλει συγγνώμη, κυρώσεις. και να αναλάβει δράση για την επικύρωση του, της ε, σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. πρέπει να γίνουν σεβαστές οι αρμοδιότητες των κρατών μελών. Η Βουλγαρία είναι ένα κράτος που έχει αρνηθεί να επικυρώσει τη σύμβαση αυτή. Είναι μια, ε, ένα ζήτημα για το οποίο έχει γίνει εκτενέστατος δημόσιος διάλογος στη χώρα μου και υπάρχει και σχετική απόφαση ανώτατου δικαστηρίου της Βουλγαρίας. Επομένως είναι ξεκάθαρο για μας ότι δεν επιθυμούμε να επικυρώσουμε αυτή τη σύμβαση και με ανησυχεί ότι κάθε φορά σε οποιοδήποτε έγγραφο συζητούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αυτή η αναφορά, αυτή η επίκληση στην σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης. Με εντυπωσιάζει αυτό, με εκπλήσει, συνάδελφοι. Όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν πρόκειται να μετακινηθούμε από τη θέση μας. Γιατί θεωρούμε ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αντίκειται στο, στις εθνικές μας παραδόσεις και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Ε, το φωνάζουμε αυτό, το διατρανώνουμε εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν φαίνεται κανείς να μας ακούει. Εμείς ε, με αυτή την τη στάση θεωρούμε ότι πειρασπιζόμαστε τις αρχές της Ένωσης, εν πάση περιπτώσει. Να σας συγχαρώ και πάρε και Λεατούμ καταφέρατε να αναδείξετε όλα αυτά τα θέματα, την ελευθερία της έκφρασης, του λόγου. Εγώ θα ήθελα όμως να ασχοληθούμε για ζητήματα που αποσχολούν ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους πολίτες και άπτονται θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ανάμεσα σε αυτά είναι το ζήτημα της μετανάστευσης και το ζητήματα των οικονομικών δικαιωμάτων. Πιο σημαντικό πιστεύω είναι να συναφερθούμε σε αυτά παρά σε αμφιλεγόμενα διεθνή κείμενα. Πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση που είχε μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησε στο Brexit. Δηλαδή, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τιμωρεί τα κράτη-μέλη της και θα τους ασκεί πολιτική πίεση όταν έχουν μια διαφορετική άποψη. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ανθίστανται σε αυτή τη φιλοσοφία. και αναφέρομαι για παράδειγμα στην πίεση που προσπαθούμε να ασκήσουμε στις κυβερνήσεις της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες διατυπώσεις, κάποιες απόψεις στο κείμενο αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Αυτή είναι η θέση του, της πολιτικής μου ομάδας ε, για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Τζαμπάσκη. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή πρέπει να απαντήσω. Δεν ζητούμε κυρώσεις, θέλουμε να ξαναδεί η Κομισιόν την εφαρμογή. Δεν πρόκειται για κυρώσεις. Σίγουρα η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να εξεταστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συζητήσουμε και σε μετέπειτα συναντήσεις, όχι τώρα, και περιμένω και τις προτάσεις σας. Άγνης Χέλλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το πρόγραμμα Erasmus ε, είναι πραγματική Euh, ε, ε, είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Ε, κάθε μέρα βλέπω και συναντώ πολλούς φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό το οποίο είναι... Α, όχι τώρα, μετά. Α, εντάξει, να τα πω μετά. Μου δώσατε το λόγο, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να μιλήσω. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ όλους. Θα έχουμε γόνιμες συζητήσεις και θα τελειώσουμε την γνωμοδότηση, αλλά υπάρχει και άλλη μια πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε. Πώς θα πείσουμε να εισακουστεί η γνωμοδότηση. Χρειάζονται λόμπι στις πολιτικές ομάδες και στη ΛΥΜΠΕ να μην το διαβάσει και το ξεχάσει το κείμενό μας. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι στις 3 το μεσημέρι στις 25 Φεβρουαρίου, που είναι αρκετά σύντομα. Και τώρα πάμε στο σημείο 7, που είναι μια αναφορά. Φτάνουμε στις αναφορές που είναι η βασική μας δουλειά η 1106 ε, του 2018 του Αλεξάνδερ Έντμπεργκ Τόρεν Σουηδικά για την έναρξη μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας εγγραφής και έγγραφο ταυτοποίησης για τους φοιτητές Εράσμου στην Ευρώπη. Ε, ο αναφέρον δεν μπορούσε να έρθει. Έχουμε τη σύνοψη και δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν Πρόκειται για την κυρία Αρνα... Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε σήμερα να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Λάβαμε τα, την ενημέρωση μέσα του 19 στην απάντηση της Κομισιόν στην αφορά εξηγούμε ότι η Κομισιόν εργάζεται πάνω στην πρωτοβουλία Ευρωπαϊκής Φοιτητικής Κάρτας που θέλει να απλουστεύσει την κινητικότητα των φοιτητών ε, σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα αυτών που αρχίζουν με το Εράσμους. Βλέπουμε ε, συνολικά το θέμα, εξυγχρονίζουμε, ψηφιοποιούμε όλες τις διαδικασίες και τις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές όταν πάνε στο εξωτερικό για σπουδές και εις επίμετρο να αναπτύσσουμε και μία, έναν ε, ηλεκτρονικό τρόπο ταυτοποίησης ώστε να μπορούν online να ε, ταυτοποιούνται όταν ζητούν διάφορες υπηρεσίες στη χώρα που τους φιλοξενεί στο ε, πανεπιστήμιο το ξένο. Επίσης θέλουμε να ενθαρρύνουμε όλα τα ιδρύματα και άλλες οργανώσεις που εκδίδουν κάρτες να ε, ενσωματώσουν στις κάρτες αυτές ένα ευρωπαϊκό ολόγραμμα ώστε να διευκολύνουμε τους φοιτητές και να αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρώπη κάρτες τους εύκολα και να έχουμε μια φοιτητική ταυτότητα που θα αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη. Όταν λοιπόν πάνε στο εξωτερικό οι φοιτητέ να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες, σε εκπτώσεις που δικαιούνται όταν είναι στο εξωτερικό. Οι αρμοδιότητες έκδοση φοιτητικών καρτών βρίσκονται στα κράτη-μέλη και ε, ε, δεν υπάρχει εναρμονισμένη διαδικασία έκδοση καρτών από τα πανεπιστήμια στα κράτη-μέλη. Οπότε δεν μπορούμε να ζητήσουμε αυτή η κάρτα η φοιτητική θα σας δίνει τη δυνατότητα να διαμένετε στην χώρα μέλος υποδοχής. Από τότε που πήραμε αυτή την αναφορά όμως, ήρθαμε σε επαφή με την ακαδημαϊκή κοινότητα και έχουμε θετικές εξελίξεις. Έχουμε το Erasmus Plus Mobile App που μπορούν έτσι να παίρνουν οι φοιτητέ όλες τις πρακτικές πληροφορίες που χρειάζονται όταν πάνε σε άλλη χώρα μέλος. Ε, αυτό έχει τώρα κατέβει πάνω από 80.000 φορές, οπότε έχουμε μια διαδικασία για τους φοιτητέ φιλική προς αυτούς και έχουμε πάνω από 2.000 ε, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που εξετάζουν τις ψηφιακές υπηρεσίες που αναπτύξαμε στα πλαίσια αυτής της ε, πρωτοβουλίας για να έχουμε απλές και εναρμονισμένες διαδικασίες για τους φοιτητές του Erasmus+. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε για να εξυγχρονίσουμε ε, ως Κομισιόν ε, τα, τις εφαρμογές και ζητούμε τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να πάνε και παραπέρα. Και τώρα έχουμε 2,3 εκατομμύρια φοιτητικές κάρτες ευρωπαϊκές που είναι έτοιμες και ενθαρρύνουμε όλα τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα να τις υιοθετήσουν. Οπότε ένας φοιτητής που σπουδάζει σε ένα πανεπιστήμιο στην Ευρώπη να μπορεί να κινείται ελεύθερα σε άλλα κράτη-μέλη ως φοιτητής για να κάνει ένα κομμάτι των σπουδών ή της εκπαίδευσής του εκεί, της ε, κατάρτισης. Ε, αυτή είναι η της εκπαιδευσης του εκει της καταρτισης αυτη ειναι η απαντηση και υπάρχουν και κάποιες ενημερώσεις τότε που λάβαμε την αναφορά. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, για τις ε, προϋποθέσεις διαμονής για τους φοιτητέ, για παραμονή πέραν των τριών μηνών, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Πανεπιστήμιο. Το κράτος μέλος της, ε, στο, στο κράτος μέλος θα πρέπει να έχει ασφαλιστική κάλυψη για να μην επιβαρύνει τα κοινωνικά συστήματα των κρατών μελών υποδοχής. Ε, σύμφωνα με την οδηγία για την ελεύθερη διακίνηση τα κράτη-μέλη είναι ε, ελεύθερα να ζητήσουν εγγραφή. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που έχουν συστήματα ε, εγγραφής, καταχώρησης των φοιτητών. Άλλοι δεν έχουν τέτοιες διαδικασίες. Αλλά για να σας ενημερώσω, αν υπάρχει διαδικασία καταχώρησης, οι φοιτητές θα πρέπει να δείξουν την ταυτότητά τους και σύμφωνα με τον κανονισμό που πέρσι εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα υπάρχουν ασφαλέστερες ε, ταυτότητες που θα κυκλοφορήσουν από την δεύτερη, Δευτέρα Αυγούστου 2020. Οπότε δεν θα υπάρχει εκεί ανάγκη ε, καταχώρησής τους στα κράτη-μέλη υποδοχής. Ευχαριστώ. Α, η Αγνές Ευρέν τώρα. Τώρα είναι η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε την Κομισιόν ε, που μας έδωσε πολύ συγκεκριμένα και ενθαρρυντικά στοιχεία. Όπως έλεγα και προηγουμένως, είναι γεγονός ότι το πρόγραμμα Erasmus Plus ε, είναι ε, πραγματικά μεγάλη επιτυχία. Την προηγούμενη χρονιά πάνω από 250.000 Ευρωπαίοι εποφελήθηκαν από αυτήν την κινητικότητα, αλλά όπως αναφέρει, γράφει και ο αναφέρον, ορισμένες να, ε, ορισμένοι νέοι μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα στην χώρα υποδοχής ε, γιατί οι διαδικασίες καταχώρησης ε, δεν αποτελούν αρμοδιότητες Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την κάθε χώρα χωριστά. Μπορώ πάντως να πω στον αναφέροντα ότι εμείς θέλουμε και απλούστευση και όπως είπε και η Κομισιόν ήδη ε, έχουν ε, προκύψει κάποιες εξελίξεις όπως ε, το Erasmus Visa Paper που έχει αποτελεί σε αντικείμενο μελέτης, δηλαδή το έχουν συμβουλευτεί πάνω από 13.000 από το ξεκίνημά του. Είναι εμβληματική αυτή η διαδικασία και θα, οπωσδήποτε θέλουμε να διατηρηθεί η χρηματοδότηση και προτείνουμε κυρία Πρόεδρε να κλείσει αυτή η αναφορά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μερίκλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Σμερίλιο. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, ε, αναφέροντα γιατί εδώ το θέμα άπτεται το της ε, ποιότητας σπουδών ε, των ε, νέων που αντιμετωπίζουν προβλήματα νομικής προστασίας αλλά και υγειονομικής κάλυψης. Η έλλειψη ψηφιοποιημένων στοιχείων μπορεί να υποβαθμίσει ε, την ε, ποιότητα των σπουδών στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το Erasmus+. Ε, για την περίοδο 2021-2027 το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συνεργάζονται στενά έτσι ώστε να ενταχθεί το, η, το ευρωπαϊκή ε, ταυτότητα ε, των φοιτητών. αυτή τη στιγμή όμως παρότι αναφέρεται στο σώμα του, του κειμένου δεν έχουμε οποιαδήποτε δεσμευτική αναφορά όσον αφορά ε, την ε, ε, ημερομηνία. Το 2021 όμως εμείς θα θέλαμε να υπάρχει αυτή η φοιτητική ταυτότητα. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα μπορεί να βελτιώσει την ε, ε, κινητικότητα των φοιτητών έστω ε, και αν η Κομισιόν θα πρέπει να βάλει και στο site του Erasmus Plus ένα ε, μια εικονική ε, ε, κάρτα την οποία θα μπορούν στην αρχή να χρησιμοποιούν οι φοιτητέ. Εγώ θεωρώ και υπό το φω των όσων ελέγχθησαν μέχρι τώρα ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά καθότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της διαδικασίας εγγραφής, καταχώρησης και ταυτότητας. Κυρίως αναφέρομαι στην καταχώρηση των φοιτητών ως κατοίκων στη χώρα υποδοχής στη διάρκεια της κινητικότητάς τους. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τις διάφορες παρεμβάσεις. Η πρόταση είναι να αφήσουμε την αναφορά ανοιχτή και να παρακολουθήσουμε ε, τις επόμενες ε, κινήσεις, γιατί υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι ασαφή προς όρασα. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 8. Ε, είναι η αναφορά 0594-2019 από τον BE, αρχικά ονόματος, γερμανικής ε, ηθαγένειας. Α, επίσης ε, αφορά την, την 841 του 2019 από την Ιταλία που αφορούν ε, την ε, ε, απαγωγή παιδιών στην Ιαπωνία. Επίσης, στην Ιαπωνία η αναφορά 842 του 2019 από τον Βενσόν Φισό από την Γαλλία, πάντα για το ίδιο θέμα, καθώς επίσης και αναφορά 843 του 2019 από την Ιταλία που αφορά το ίδιο θέμα απαγωγή παιδιών από την Ιαπωνία. Έχουμε εδώ τους αναφέροντες. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να έρθετε στις Βρυξέλλες. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε λοιπόν. Δεν ξέρω BE από την Γερμανία είναι τα αρχικά σας. Έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά ο καθένας. Σας ευχαριστώ. Θα μοιραστώ το χρόνο με τον πρόεδρο της οργάνωσης ε, για τα παιδιά που έχει έρθει μαζί μου από την Γαλλία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε να αναδείξουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο προκαλεί ψυχολογική και προβλήματα σε παιδιά που είναι αδύνατα να εκφράσουν εκείνα τη θέση τους. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τις επιπτώσεις της αρπαγής ανηλίκων. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη Σύμβαση της Χάγης για την πρόληψη της διεθνούς αρπαγής ανηλίκων. Έχω εγώ εδώ τα διαβατήρια των παιδιών μου, Καρλ Λιώχαν. Η πρώην σύζυγός μου έχει ε, προβλήματα ε, προσωπικότητας, ψυχολογικά και δεν τα έχω δει τα παιδιά εδώ και 11 μήνες έχουμε προσπαθήσει τρεις φορές ε, να γίνει έμεση ε, εφαρμογή της δικαστικής απόφασης που θα έδινε σε εμένα την ε, πατρότητα, αλλά αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό. Και... και επιδιώκουμε τον επαναπατρισμό τους. δεν, δεν έχω, δεν είχα καμιά επικοινωνία μαζί τους μέχρι στιγμής. Έχει κινητοποιηθεί και το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Υπάρχει επίσης απόφαση Ιαπωνικού δικαστηρίου α, στην περίπτωση του Βίλεμ. Εάν και έχει δοθεί στον γονέα αυτόν μια απόφαση δικαστηρίου που του δίνει πολλές, ε, ε, τη δυνατότητα να επισκέπτεται τα παιδιά του σε μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχει εφαρμοστεί. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Το Μάσκη Κατερίνα. Αρπαγή ανηλίκων στην Ιαπωνία. Πρόκειται δηλαδή για εσωτερική υπόθεση, όχι για διεθνή. Και πάλι όμως δεν μπορεί το παιδί για δυόμιση χρόνια να δει τον πατέρα του. Και επίσης έχουμε πολλούς γονείς που επικοινωνούν μαζί μας και μας λένε ότι φοβούνται, ότι μπορεί να απαγάγει τα παιδιά ή σύζυγός τους και να μην τα ξαναδούν ποτέ. Εγώ τρία χρόνια προσπαθώ να αντιμετωπίσω αυτή την αρπαγή των παιδιών μου στην Ιαπωνία και πάνω από χίλια παιδιά έχουν αρπαγεί από την Ευρώπη προ την Ιαπωνία από το τέλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα. Πάνω από χίλια παιδιά. Κάτι πρέπει να κάνουμε για όλο αυτό το θέμα. Είμαι πρόεδρο τη γαλλική οργάνωση Αλόν Λεζονφών. Και έχω εργαστεί και ω διερμηνέα Ιαπωνικών για τα γαλλικά δικαστήρια. Η συζήτηση σήμερα αφορά τα δικαιώματα χιλιάδων γονέων. Μια χώρα η οποία παραβιάζει τα θεμελιώδη τους δικαιώματα να έχουν πρόσβαση στα παιδιά τους. Στην Ιαπωνία δίνεται πλήρης δυνατότητα, στο, στο, ε, ε, δικαιώματα στον γονέα που έχει μείνει πίσω. Και δεν δίνεται δυνατότητα επίσκεψης στον άλλο γονέα. Το 2014 επικύρωσε τη Σύμβαση της Χάγης η Ιαπωνία, όμως αμέσως μετά οργανώθηκε σεμινάριο στο Παρίσι από τις Ιαπωνικές Αρχές για να ενημερώσουν ουσιαστικά τους πολίτες τους που ζούσαν στο Παρίσι πώς μπορούν να νομιμοποιήσουν μια αρπαγή ανηλίκου τώρα που ετέθησε εφαρμογή η Σύμβαση της Χάγης. ακόμα και αν ο γονέας είναι ο μόνος, που έχει, ο επιζών και ζει στην Ιαπωνία, πάλι δεν θα έχει πρόσβαση στο παιδί του. Είχαμε μια υπόθεση, ένα παιδί που έχει απαχθεί πριν από τρεις εβδομάδες. Δεν θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε αυτό οι γονείς του, γιατί γιατί χρειάζεται επιστολή από τη σύζυγό του ο πατέρας για να πάρει βίζα θεώρηση για να το επισκεφτεί στην Ιαπωνία. Μετά δηλαδή από ένα εξαναγκαστικό διαζύγιο στην Ιαπωνία και από την πλήρη στέρηση των δικαιωμάτων του, ε, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και έχουμε αντίστοιχες περιπτώσεις από γονείς που έρχονται από πολλές άλλες χώρες, από την Αμερική, από την Αυστραλία, από τον Καναδά και άλλες. Ευχαριστώ. Οι, όλοι οι αναφέροντες, ο Πολ Ζορστούγια, α όχι εσείς, εσείς μιλήσατε ήδη, με συγχωρείτε, συναναφέρον. Βενσάν Φυσό. Έχετε το λόγο. First of all, let me... Uh, Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τα μέλη του Κοινοβουλίου, την Κομισιόν, ιδιαίτερα τον Ινιάσο Κοράο, αλλά και Γάλλους βουλευτές που δραστηριοποιήθηκαν υπέρ ημών και των παιδιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Βενσάν Φυσό. Τα παιδιά μου απήχθησαν πριν από 559 ημέρες έχουν και γαλλική υπηκότητα. Την τελευταία φορά που είδα την κόρη μου ε, ήταν ε, από ένα σύστημα κλειστής τηλεόρασης, κλειστού κυκλώματος, ήταν 11 μηνών, ήταν καλοκαίρι και έφευγαν ε, μέσα, στο, μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ε, πήγα στο Τόκιο τέσσερις φορές, ε, κατήγγυλα, ε, κακή, κακοποίηση, απαγωγή, υπό αστυνομία αρνήθηκε να με βοηθήσει και όταν τους είπα ότι θα πάω να βρω τα παιδιά μου μόνος μου, η παρουσία δικηγόρου με κατηγόρησαν, μου άφησαν κατηγορίες. Ε, ζήτησα να την εξετάσουν ε, ειδικοί να εξετάσουν και τα παιδιά. Το γαλλικό προξενείο στο Τόκιο προσπαθεί πάρα πολύ να βοηθήσει τα παιδιά ε, και πολλές φορές κάλεσε την ε, γυναίκα μου για να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι εν ζωή. Κάθε φορά απέτυχε. Οι Ιαπωνικές αρχές δεν έκαναν τίποτα και δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο τις γαλλικές αρχές να βρουν που είναι τα παιδιά μου, τα απαχθέντα το κράτος δικαίου δεν εφαρμόζεται σε αυτή τη χώρα. Κάναμε αναφορά στον ΟΗΕ κατά της Ιαπωνίας, τέλος του περασμένου έτους. Και καταδείξαμε ότι η Ιαπωνία δεν σέβεται την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Για να δείξω την υποκρισία των Ιαπωνικών αρχών, θέλω να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Στις 21 Νοεμβρίου, ο Ιάπων πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη είπε ότι για τον εορτασμό των 25 ετών τη κύρωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Παιδιών δεσμευόταν η Ιαπωνία να υλοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις. Ε, δυο, μια μέρα μετά είπαν ότι η σύμβαση δεν έχει δεσμευτική ισχύ στην Ιαπωνία. Έχει διπλή γλώσσα η Ιαπωνία. Ε, λέει ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα για να ε, ε, προσχωρήσει σε λέσχες των ισχυρών αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνουν τίποτα λένε ψέματα στους εμπορικούς εταίρους και στους συμμάχους τους το ψυχολογικός αντίκτυπος είναι σοβαρός για τα παιδιά μας πολλές μελέτες δείχνουν την μακροπρόθεση, το μακροπρόθεσμα αντίκτυπο σωματικό και ψυχολογικό όλων αυτών στα παιδιά. Ε, αυτό ταξινομείται και ως νόσος. Ε, όταν ζητούμε από την Ιαπωνία να εξεταστούν από ειδικό τα παιδιά, απορρίπτεται το αίτημα. Ε, είναι σαν να έχει κάποιος καρκίνο και να αρνούνται να κάνουν την εξέταση και τη διάγνωση οι ειδικοί. Τα παιδιά πρέπει να γυρίσουν πίσω σε ένα περιβάλλον που θα τα φροντίσει, που θα σέβεται τα καλύτερα συμφέροντά τους να μένουν μαζί με τους γονείς ε, που δεν πρέπει να αποξενώνονται. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, σωστά σωματικά και ψυχολογικά. Τα παιδιά μας έχουν αποξενωθεί από την Ευρώπη. Δεν μιλάνε πια τη γλώσσα μας, δεν έχουν τη θρησκεία μας. Δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν στη χώρα καταγωγή τους για να επισκεφτούν τον πατέρα τους που μπορεί να πεθαίνει. Πώς δεν γίνει αποδεκτό αυτό. Η ολοκλήρωση είναι ο πυλώνας της κουλτούρας μας στην Ευρώπη. Ένα μη Ευρωπαίος ε, έρθει στην Ευρώπη, κάνουμε ό,τι δυνατόν για να διατηρήσει την πολιτιστική του ταυτότητα. Αυτή η Επιτροπή πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εφαρμοστούν τα ίδια δικαιώματα ε, για τα παιδιά μα εκ των συνόρων, ιδιαίτερα σε μια χώρα η οποία αποκαλεί τον εαυτό τη φίλο τη Ευρώπη. Εν ώψη της κακής πίστης της Ιαπωνίας και παρά τις πολλές προσπάθειες Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης να φροντίσουν ώστε τα παιδιά μας να έχουν τα δικαιώματά του σεβαστά, ε, η Ιαπωνία κοφεύει. Έτσι ζητούμε κυρώσεις. Ε, εδώ και χρόνια, για να μην σας πω δεκαετίες, προσπαθούμε με την Ιαπωνία και μας λένε ψέματα κατάμουτρα. Ε, και ο υπουργό των Εξωτερικών είπε ότι δεν θα εφαρμόσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε κυρώσεις εναντίον τους. Δεν είναι ψέματα και εδώ καλούμε άμεση αναστολή της ε, Συμφωνίας ε, Στρατηγικής ε, Εταιρικής Σχέσης. Εστάλουν τις ανεπιστολές στους Υπουργούς της Ιαπωνίας για την, το σεβασμό της Σύμβασης για τα δικαιώματα των παιδιών. Η Ιαπωνία δεν σέβεται το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λίγους μήνες αργότερα μετά από αυτό η Ευρώπη υπέγραψε τη Συμφωνία εταιρική Σχέσης. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Η δεύτερη κύρωση είναι άμεση ε, ε, ε, εισαγωγή υποχρέωση θεώρησης για τους Ιάπωνες που έρχονται εδώ. Δεν μπορεί ατιμωρητοί να αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας έτσι. Πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα στην Ιαπωνία ότι αυτά τα εγκλήματα δεν θα πάνε, περάσουν ατιμόρυτα. Τέλος, μετά το παράδειγμα της Ιταλίας, να καλέσουμε τα κράτη-μέλη που ε, έχουν ε, παρουσία στην Ιαπωνία να ενημερώσουν τους πολίτες τους για τον κίνδυνο απαγωγής εάν επισκεφθούν ή διαμείνουν στην Ιαπωνία. Δεν πρέπει άλλα παιδιά να απαχθούν. Αν είχαν ληφθεί τα μέτρα αυτά πριν από χρόνια, τα παιδιά μας δεν θα είχαν απαχθεί. Είναι ο καιρός για δράση. Τελειώνοντας, να πω ότι πολλές φορές οι νομοθέτες μου λένε ότι είναι κυρίαρχο Κράτο ή η Ιαπωνία, αλλά και η Ευρώπη είναι όταν πρόκειται να αποφασίσει τη φύση οικονομικών και διπλωματικών σχέσεών της με την Ιαπωνία. Θα πρέπει να ε, ε κινηθούμε. Δεν μπορεί να μην χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και να αφήσουμε την Ιαπωνία να κινείται ε, τελείως ε, ασίδωτα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε την ιστορία, τις ιστορίες σας μαζί μας. Είστε τέσσερις, επομένως αν θέλετε παρακαλώ να πάρετε το λόγο. Ε, πέτε μας ε, ποιος είστε, γιατί δεν σας έχω τον... Η 841 είναι η δικιά μου. Ε, λέγομαι Τομάζο Περίνα, Ιταλική, Ιταλός ε, υπήκος και ε, το 2003 ξεάρχισα να δουλεύω στην Ιαπωνία. Τον, από το Δεκέμβριο του 2016 μέχρι το 2019 δεν ε, έζησαν με την μητέρα τους και έχω χίλιες μέρες που δεν τα έχω δει. Είμαι ακόμα παντρεμένος ε, με την ε, γυναίκα μου. Δεν έχω κανένα είδος περιορισμού πρόσβασης στα παιδιά, μας, παιδιά μου. θα είχα όλα τα δικαιώματα να επισκέπτονται με τα παιδιά μου εάν ζούσα σε μια, οικογέ... σε μια χώρα που σέβεται τα δημοκρατικά δικαιώματα. Ε, τα ανώτερα δικαστήρια, το ειδικό δικαστήρια, ε, όλα έχουν ε, ό,τι έκανα όμως δεν είχε αποτέλεσμα. Το παιδιά μου μαζί με πολλά άλλα παιδιά. Ε, ε, δεν πρόκειται να τα δώσει η Ιαπωνία. Διεφθαρμένο δικαστικό σύστημα και ένα σωρό άλλα προβλήματα μου εμποδίζουν να δω τα παιδιά μου. Ε, δεν μου δίνουν δίκιο ούτε οι υπόλοιπε δημόσιες αρχές. Η αστυνομία είπε ότι ε, ε, ε, στην αστυνομία που στράφηκα είπε ότι θα ασχοληθεί με το θέμα, αλλά στην ουσία ένα χαστούκι παραπάνω δέχτηκα γιατί μου είπαν ότι στην Ιαπωνία δεν είναι παράνομο να απαχθεί ένα παιδί από τους γονείς του. Το Ιταλικό προξενείο έκανε προσπάθειες και να έρθει σε επαφή με την αστυνομία και την σύζυγό μου επανειλημμένα. Ωστόσο η Ιαπωνία δεν απήντησε ούτε μία φορά παραβιάζοντας ε, τη συνθήκη της ε, Βιέννης. Το 2018, τον Οκτώβρη, ο Λορέντζο Φοντάνα, ε, υπουργό ε, για θέματα οικογένειας, έγραψε στο μόλογό του να μάστα ε, για το θέμα αυτό. Μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Επίσης, ο Σέντζο Ματαρέλα, πρόεδρος της Ιταλίας, όταν ο Ιάπωνα Πρωθυπουργό επισκέφθηκε την Ιταλία, αναφέρθηκε στον προβληματισμό αυτό χωρίς να λάβει καμία απάντηση. Επίσης, ε, και άλλος αρμόδιος υπουργός ε, ε, σε επίσκεψή του στην Ιαπωνία ήγηρε το θέμα αυτό χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ο Τζουζέπε Κόντε στην Οζάκα στη διάρκεια της συνεδρίασης του G20 αναφέρθηκε στην τραγική κατάσταση των απαχθέντων παιδιών ε, αλλά ο Πρωθυπουργό Άμπε είπε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι γιατί δεν μπορεί να επηρεάσει τους δικαστές του. Την, το προηγούμενο Νοέμβριο η Μάρα Καρφάνια ε, σε επίσκεψη στην Ιταλία ε, ως πρόεδρος της Βουλής μίλησε στον ομόλογό της για το θέμα των παιδιών Ιταλών υπηκών για μία ακόμα φορά χωρίς αποτέλεσμα. Ε, η προξενική προστασία βάσει της συμβάσεως της Βιέννης ε, δεν γίνεται σωστή, δεν γίνεται σεβαστή ε, και τα παιδιά μας εν τέλει δεν έχουν δικαιώματα σε μια χώρα που υποτίθεται ότι είναι σύμμαχος και φίλοι. Επίσης, οποτεδήποτε προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε τα δικαιώματά μας, ε, στην ουσία μας απείλησαν ε, το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Προστασία των, παιδιών, των Δικαιωμάτων των Παιδιών CSC, ε, καθώς, CRC, καθώς επίσης και το άρθρο 35 της Ιδίας Συμβάσεως παραβιάζονται διαρκώς η Ιαπωνική κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να σεβαστεί ε, την συμφωνία, την σύμβαση CRC και δείχνει η κυβέρνηση της Ιαπωνίας πάντα πολύ κακή πίστη δεν έγιναν ε, σεβαστά τα δικαιώματα επίσκεψης που έχω, αλλά χωρίς καμία ε, ε, ποινή. Τα παιδιά Ευρωπαίων πολιτών δεν έχουν δικαιώματα, δεν μπορούν να μιλήσουν τη γλώσσα τους, δεν μπορούν να μιλήσουν με την μισή τους οικογένεια, δεν μπορούν να μάθουν την μισή τους κουλτούρα. Αυτά τα παιδιά έχουν πάψει να είναι παιδιά από την Ευρώπη. Δεν έχουν ε, ε, καμία συνέχεια πολιτιστική και δεν γνωρίζουν την πολιτιστική τους κληρονομιά. Αυτά δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν. Ε, η, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα γνωρίζει αυτά. Παρ' όλα αυτά έχει υπογράψει συμφωνία εταιρική σχέσης ε, και συμφωνία οικονομικής εταιρική σχέσης με την Ιαπωνία. Επομένως, εδώ προτίθεται το ερώτημα. Από τη στιγμή που εξακολουθούν πολλά παιδιά να μην έχουν δικαιώματα στην Ιαπωνία, μα ενδιαφέρει, ενδιαφέρει μόνο η οικονομία και το εμπόριο ή και τα παιδιά. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν άμεσες κυρώσεις ε, κατά της κυβέρνησης της ε, Ιαπωνίας. Εάν τα μέτρα αυτά είχαν ληφθεί μερικά χρόνια πριν, δεν θα είχαν υποστεί αυτά τα εγκλήματα, τα φρικαλέα, τα παιδιά μας. Τρία πράγματα ζητούμε. Ζητούμε να σταματήσει αμέσως η συμφωνία SPA επίσης ε, να ε, υπογράψουν ε, κοινή επιστολή οι πρέσβεις στην οποία θα αναφέρουν προς την Ιαπωνική, μάλλον έγινε μια τέτοια επιστολή από τους πρέσβεις, δεν υπήρξε καμία απάντηση από Ιαπωνική πλευρά. αντιθέτως μερικούς μήνες μετά το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη Συμφωνία SPA. Ε, ζητούμε να δυσκολευτεί το ταξίδι των Ιαπώνων ή στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και επίσης η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στο Τόκιο ε, και οι λοιπές αρχές να εκδίδουν οδηγίες προς τους ταξιδιώτες για τα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν. Ε, κακή πίστη, ε, ακινησία έδειξε η Ιαπωνική κυβέρνηση. Εμείς βρισκόμαστε σε απόγνωση και σας παρακαλούμε να μας βοηθήσετε για να ξαναδούμε τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, η Γραμματεία... Έχουμε εκπρόσωπο της Κροατικής Προεδρίας με ενημερώνει η Γραμματεία. Βέβαια θα ακούσουμε πρώτα την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Πατρίθια, Ντελούκα, είστε εδώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να εκφράσει την κατανόηση της για την ε, δύσκολη ε, κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι αναφέροντες. Γνωρίζουμε την κατάσταση στην Ιαπωνία και όσον αφορά την επιστροφή ενός ανηλίκου μετά την αρπαγή του στην συνήθη κατοικία του, καθώς επίσης και τις δυσχέρειες που υπάρχουν στην άσκηση των δικαιωμάτων επίσκεψης. Ακόμα και όταν αυτά τα δικαιώματα επίσκεψης έχουν αναγνωριστεί από δικαστήριο. Επίσης συμφωνούμε ότι δεν εφαρμόζεται ε, δεν υπάρχει μάλλον σύστημα κοινή επιμέλεια, ότι μόνο σε ένα από τα μέρη δίνεται επιμέλεια στην Ιαπωνία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα και για του Ιάπωνες πολίτε. Για παράδειγμα, εάν έχουμε ε, την επιμέλεια να έχει δοθεί στη γυναίκα και αυτή ξαναπαντρευτεί, δίνεται η δυνατότητα να υιοθετηθεί από τον νέο σύζυγο το παιδί, χωρίς καν να ενημερωθεί ο φυσικός γονέας του παιδιού. Αυτό είναι απίστευτο, θα ήταν αδιανόητο στο δικό μας νομικό πολιτισμό. Αλλά δυστυχώς εδώ πρέπει να γίνει σεβαστή η αρχή της μη ε, επέμβασης. Γιατί ουσιαστικά το αστικό δίκαιο στην Ιαπωνία θεωρεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι αμυγός ιδιωτικής φύσεως και ότι το κράτος δεν θα πρέπει να επεμβαίνει. Αυτή είναι η νομική τους φιλοσοφία. Το αποτέλεσμα είναι αδυναμία επιβολής των δικαστικών αποφάσεων σε τέτοια αστικά ζητήματα. Έχουν αναλυφθεί πολλές πρωτοβουλίες για να υπάρξει ευαισθητοποίηση των Ιαπωνικών αρχών, να τους επισημάνουμε το πρόβλημα. Οι αναφέροντες ανέφεραν ορισμένε από αυτές τις ε, πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα την επιστολή των 26 πρέσβεων. Και βέβαια έχουν υπάρξει παρεμβάσεις και σε πολιτικό επίπεδο. Μετά την επιστολή τον πρέσβεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Γιούροβα, πρώην Επίτροπος Δικαιοσύνης, είχε αποστείλει επιστολή στον ομόλογό της, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Καμικάβα. Βέβαια δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Επίσης, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τόκιο έχει επιδιώξει συνάντηση με τον Υπουργό Τακάση Γιαμασίτα το 2019, το επεδίωκε, και με εκπροσώπηση όλων των πρέσβεων των κρατών μελών στο Τόκιο. Αυτή η συνάντηση δεν έγινε ποτέ. Ο Υπουργό ε, της Ιαπωνίας, ωστόσο, συναντήθηκε με τον επικεφαλής της, εκπροσω... της αντιπροσωπείας της Ένωσης στο Τόκιο. Είχε σημασία αυτή η συνάντηση για να συνεχίσει να είναι ανοιχτό το... ανοιχτός ο διάβλος της επικοινωνίας, αλλά δεν βγήκε τίποτα ουσιαστικό τον Ιούνιο του 2019 ο Γάλλος πρόεδρος ο κ. Μακρό και ο κ. Ντεκόντε ε, της Ιταλίας και άλλοι ε, έκαναν επαφές και παρεμβάσεις προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιαπωνίας, αλλά δεν συνέβη τίποτα. Ο κύριος Μασάκο Μόρι είναι ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης της Ιαπωνίας από τον Οκτώβριο και μετά θα επιδιώξουμε επικοινωνία μαζί της για να δούμε εάν θα είναι πιο ανοιχτή προς τη συζήτηση αυτών των θεμάτων σε σχέση με τους συναδέλφου τη. Μετά από όλη αυτή τη διεθνή πίεση, γιατί γνωρίζετε ότι και άλλες, χώρε χώρες, αναφέρατε τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, έχουν αντίστοιχα προβλήματα, υιοθέτησε νέα νομοθεσία η Ιαπωνία, ε, την ε, πράξη για την εφαρμογή ε, αστικών αποφάσεων αστικού δικαίου. Όμως, ε, αμφιβάλλουμε για το κατά πόσον θα εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία και πόσο αποτελεσματική θα είναι. Δεν έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμογή. Θα τεθεί σε εφαρμογή τον Απρίλιο του 20. Αναφέρετε και εσείς τη Στρατηγική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης. 31 Ιανουαρίου έγινε η δεύτερη συνάντηση στο πλαίσιο αυτής της ε, στρατηγικής σχέσης με τις αρχές της Ιαπωνίας. Βέβαια πρέπει να επιθυμήσω ότι η Συμφωνία Στρατηγικής Σχέσης δεν έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμογή γιατί δεν έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, κάποια στοιχεία της ε, συμφωνίας εφαρμόζονται σε προκαταρκτικό επίπεδο. Δεν εφαρμόζεται όμως το σκέλος της συμφωνίας που αναφέρεται στη συνεργασία στο αστικό δίκαιο, όμως τα ε, διατάξεις της συμφωνίας που αφορούν στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εφαρμόζονται ήδη. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτών ζητήσαμε εξηγήσει για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το νέο σύστημα διεθνούς μεσολάβησης που προωθεί η Ιαπωνία. Ζητήσαμε επίσης στατιστικά στοιχεία πόσα είναι τα παιδιά που μπόρεσαν να επιστρέψουν στην, στον συνήθι τοποκατοικία τους, μετά από αρπαγή. Τα ζητήσαμε αυτά από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας. Δεν λάβαμε ικανοποιητικέ απαντήσεις, πρέπει να σας πω. Αλλά θα γίνουν άλλες δύο ε, συναντήσεις για, στο πλαίσιο του διαλόγου που κάνουμε για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μετά προβλέπεται και η Σύνοδος Κορυφής στο Τόκιο το Μάιο. Τα θέματα λοιπόν αυτά θα συνεχίσουμε να τα θέτουμε, επιδιώκοντας να λάβουμε μια συγκεκριμένη απάντηση. Την 25η λοιπόν επέτειο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εορτάσαμε φέτος, και πάλι η αντιπροσωπεία της Ένωσης στο Τόκιο προσπάθησε να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα θέματα αυτά. Προσπαθήσαμε να δημοσιοποιήσουμε άρθρα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στην Ιαπωνία. Αλλά όπως έλεγα είναι ένα πρόβλημα στο οποίο συμπλέκονται πολλά. Πρέπει να γίνουν σεβαστές διεθνείς συνθήκες όπως η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αλλά επίσης διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν βασικές πολιτιστικές διαφορές. Γιατί εμείς οι Ευρωπαίοι αντιλαμβανόμαστε ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού είναι ότι ακόμα και μετά από ένα διαζύγιο να έχει, την, να έχει επικοινωνία και με τους δυο γονείς του. Με άλλα λόγια, επιδιώκουμε, ε, ε, ε, μάλλον, ενώ εκείνοι θεωρούν ότι για να μπορέσει το παιδί να συνεχίσει τη ζωή του θα πρέπει να μην το ενοχλεί ο πατέρα εκείνο στον οποίο δεν δόθη η επιμέλεια. Αυτή είναι η δική του φιλοσοφία. Προσπαθούμε λοιπόν να συνεχίσουμε το διάλογο και την επικοινωνία με τι Ιαπωνικέ αρχέ. Έχουμε κάνει όλα τα απαιτούμενα διαβήματα ε, σε διπλωματικό επίπεδο και προσπαθούμε να συνεργαστούμε και με άλλα κράτη με τα οποία έχουμε παρόμοια αντίληψη όπως τις Ηνωμένε Πολιτείε για να συνεχίσουμε να θέτουμε το θέμα αυτό στις Ιαπωνικές αρχές. Τώρα σε σχέση με τις κυρώσεις. Είναι ένα θέμα για το οποίο δεν μπορώ εγώ να απαντήσω. Η επιβολή κυρώσεων προς μια τρίτη χώρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να εγκριθεί στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με ομοφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τώρα, η Ευρωπαία Συντονίστρια για τα Δικαιώματα των Παιδιών, η κυρία Εύα Κόπατς. Χάρη ε, σε εκείνη ε, πάντοτε ε, το Κοινοβούλιο εργάζεται υπέρ των βέλτιστων συμφερόντων των παιδιών. Η κυρία Κόπατς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω πολωνικά. Κυρίες και κύριοι, αυτά που ακούσαμε δηλώνουν ότι οι γονείς τα τελευταία χρόνια ζούνε απελπισμένοι. Δεν υπάρχουν ανοιχτοί δρόμοι πολύ μπροστά τους, έχουν κάποια δικαιώματα με βάση τους ευρωπαϊκούς κώδικες αλλά και τον Ιαπωνικό που όμως πολλές φορές δεν έχει εφαρμοστεί ή τύχει σεβασμού στην Ιαπωνία. Όλοι μας φανταζόμαστε τη δύσκολη κατάσταση πώς να ζήσεις χωρίς να βλέπεις τα παιδιά σου, χωρίς να ξέρεις που είναι, τι κάνουν, αν είναι καλά, αν όχι. Κάποιοι αναφέροντες που έχουμε μαζί μας το 2018 υπέβαλαν τις πρώτες αναφορές, οι αιτήματα στο γραφείο του συντονιστή και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί αυτές οι περιπτώσεις δεν ε, επιλήθησαν μέχρι τώρα παρόλο που έγιναν πολλές ε, παρεμβάσεις πολλές φορές σε ανώτατο διπλωματικό επίπεδο. Σήμερα έχουμε πολύ συγκεκριμένες αναφορές μπροστά μας. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μόνο αυτές οι αναφορές, γιατί το πρόβλημα είναι συστημικό, το οποίο προέρχεται από νομικά προβλήματα και την ιαπωνική κουλτούρα. Η κοινή επιμέλεια ε, μετά το διαζύγιο δεν προβλέπεται. Επίσης ε, δεν είναι εύκολο να ασκηθούν τα δικαιώματα επισκέψεων. Αυτό βλάπτει το ίδιο το παιδί πρωτίστως. Το παιδί χάνει όχι μόνο τον άλλο γονέα, χάνει επαφή με, μια ολόκληρη κουλτούρα, μια γλώσσα που είναι κομμάτι του κουλτούρας του. Οι γονείς σε όλο τον κόσμο, στην Ένωση, στην Αμερική, την Αυστραλία, αλλά και οι ίδιοι οι Άπωνες πρέπει να αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα μετά το διαζύγιο από τον Ιάπωνα συντροφό ή την Ιαπωνίδα ε, χάνεται η επαφή με τα παιδιά πολλές φορές σχεδόν ολοκληρωτικά ως υπεύθυνη για τα δικαιώματα του, των παιδιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζω τα εξής πάντοτε θα καταγγέλω τον μη σεβασμό δικαιωμάτων παιδιών σε οποιοδήποτε κράτος. Αυτά τα δικαιώματα υπάρχουν στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Δεν έχει σημασία αν είναι κράτος μέλος της Ένωσης ή άλλο κράτος. Ε, εδώ δοκιμάζεται η δημοκρατία, ο πολιτισμός κάθε χώρας. Θα πρέπει να καλύπτονται τα υποθέσεις αυτές. Οι όταν διακυβεύεται η καλή κατάσταση του παιδιού έχει το δικαίωμα να έχει επαφή για να διασφαλίζει ότι αναπτύσσεται σχέση γονέα παιδιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε παιδί, όχι μόνο για τα μικρά παιδιά αλλά και για τους εφήβους. Και επίσης ε, συνεχίζεται η σχέση όταν ο έφηβος θα γίνει ενήλικος. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε αλλαγές στο Ιαπωνικό δίκαιο που θα γίνουν σε λίγους μήνες και που θα επιτρέψουν επιτέλους την, τον επαναπατρισμό μετά την απαγωγή. Θα είναι αποτελεσματικές αυτές οι αλλαγές. Αυτό είναι το ερώτημα. Δυστυχώς ακούσαμε εμπειρογνώμονες να αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των νέων ρυθμίσεων. Όμως πιστεύω ότι ο διάλογος είναι πολύ σημαντικός και γι' αυτό οποιαδήποτε θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις των γονέων θα πρέπει να είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξή μας και όταν πρόκειται για ανταλλαγές απόψεων με οποιασδήποτε αρχές από την Ιαπωνία. Εγώ μίλησα με εκπροσώπους από την Αντιπροσωπεία Ένωσης Ιαπωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι το θέμα αυτό θα είναι πολύ ε, γνωστό, θα το ξέρουν τα μέλη στην επόμενη διακοινοβουλευτική συνάντηση της αντιπροσωπείας της Ένωσης και της Ιαπωνίας αυτό το θέμα θα θίγει. Επίσης, με αυτή την ευκαιρία μίλησα με τον, με, εκπρόσωπο της Ένωσης για την ασφάλεια και εξωτερικά θέματα, γιατί θέλω το θέμα αυτό να αναφερθεί κατά τις συνομιλίες που διεξάγονται τώρα, προκειμένου περί της νέας στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία. Γνωρίζω ότι οι Γάλλοι ε, σε ανώτατο επίπεδο μίλησαν με τους Ιάπωνες ομολογούς τους για το ίδιο θέμα. Κυρίες και κύριοι, οι επαφές όταν πρόκειται για γονεϊκά θέματα, οικογενειακά θέματα, κυρίως όταν πρόκειται για απαγωγές τέκνων ή επιμέλεια μετά από διαζύγιο, αυτά τα θέματα είναι από τα σημαντικότερα καθήκοντα ε, με τα οποία ασχολείται το γραφείο μου. Γι' αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Είναι η πρώτη συνάντηση όπου μιλώ συντονίστρια. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών. Θέλω να πω ότι ελπίζω ότι δεν θα χρειάζεται να συναντώμεθα πολύ συχνά γιατί δεν θα υπάρχουν πολλά περιστατικά που αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών, αν και ξέρω ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Είναι πάρα πολλές οι αναφορές που στέλνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφορούν αυτό το θέμα. Επίσης, ε, εκφράζω ε, όλη μου τη συμπάθεια προς τους αναφέροντες ε, μετά από τις επιστολές που εστάλησαν. Πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά που ζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης, συνεργασία σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε διοικητικό επίπεδο προκειμένου περί των δικαιωμάτων των παιδιών. Επί τη βάση της απόφασης του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ως μέλη της Επιτροπής και ως αναφέροντες ότι είμαι στη διάθεσή σας προκειμένου περί συνεργασίας επί αυτών των θεμάτων. Ελπίζω ότι οι επόμενοι μήνες θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών για τα πολύ δύσκολα αυτά θέματα. Η πόρτα στο γραφείο μου παραμένει ανοιχτή για τον καθένα σας, για όλους όσους θέλουν να μιλήσουν για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Κόπιτς. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος από τα μέλη θέλει να πάρει το λόγο. Αλλιώς θα πάρω εγώ το λόγο. Α, ναι. Ωραία, παρακαλώ. Ε, ε, ε, είναι απίστευτα αυτά που άκουσα. Εντάξει, όλοι έχουμε ακούσει διάφορα σε ιστορικά βιβλία τι έγινε ας πούμε το 17ο αιώνα που δεν μπορούσαν να φύγουν. forever. But I could never imagine that it can happen. μισθοφόροι δεν, στο Ναγκασάκι δεν μπορούσαν να επισκεφθούν συγκεκριμένα μέρη της ε, πόλης κλπ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα εδώ ακούμε πράγματα απίστευτα. Και βλέπουμε ότι και διάφορα διαβήματα έχουν οδηγήσει σε ε, μηδενικά αποτελέσματα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει ε, να συζητήσουμε το θέμα ε, αυτό δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται ισχυρή θέση του εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλές ε, κυβερνήσεις από ό,τι φαίνεται έχουν ε, ασχοληθεί με το θέμα, κυβερνήσεις, ε, υπότος εκπρόσωπος, πρόεδρε κτλ. Αλλά θα πρέπει κάπως η θέση να γίνει πιο ισχυρή από το Κοινοβούλιο. Μια άλλη πρόταση βεβαίως θα είναι να καλέσουμε τον ύπατο εκπρόσωπο για τις εξωτερικές υποθέσεις να έρθει εδώ να μιλήσει ε, ενώπιόν μας. Παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει το λόγο τώρα. Εγώ να μιλήσω πρώτος, λέει ο κύριος Κοράο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς καταγγείλαμε αυτό την προβληματική κατάσταση και ανησυχητική κατάσταση ε, που απειλεί παιδιά ε, Ευρωπαίων πολιτών στην Ιαπωνία, αλλά δεν είδαμε ε, καμία βελτίωση. Ο Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας ανέφερε ότι το 2020 θα είναι μια σημαντική χρονιά για τις διεθνείς σχέσεις ε, της Ιαπωνία, Ωστόσο τίποτε δεν έγινε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την κατάσταση που εξακολουθεί να υπάρχει ε, πάνω από 100 ε, παιδιά Γάλλων υπηκών και πάνω από 1000 παιδιά στο σύνολο Ευρωπαίων πολιτών παραμένουν ε, εγκλωβισμένα. Ο κύριος Τομάζο ήρθε σε επαφή μαζί μου και ανέφερε το, αυτές τις τρομακτικές ε, ιστορίες που ακούσαμε και εδώ τι πρέπει να κάνουμε, ενδεχομένως ε, να, να μετανιώσουμε που υπογράψαμε τη συμφωνία για την Ισπανία. Ίσως να ζητήσουμε από την Κομισιόν ε, να αναθεωρήσουν την ε, συμφωνίες SPA και EPA λόγω παραβίασης της ερήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά, τα δικαιώματα των παιδιών. Ίσως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με την Ιαπωνία, ε, να πιέζουμε διαρκώς την Ιαπωνική κυβέρνηση ε, και να κάνουμε τη φωνή μας ε, ισχυρή έτσι ώστε να καταλάβουν ότι διαφορετικά θα έχουν να υποστούν οικονομικές κυρώσεις. Αυτή τη χρονιά οργανώνονται το καλοκαίρι Ολυμπιακοί και Παραλυμπιακοί αγώνες ε, εκατομμύρια άνθρωποι θα στραφούν προς την Ιαπωνία. Πιστεύω ότι εδώ μπορούμε να βρούμε ένα ε, εργαλείο πίεσης, ε, πίεσης επί των Ιαπωνικών αρχών. Ε, υπάρχουν άνθρωποι στην Ιταλία, στην Γαλλία, στη Γερμανία που περιμένουν αναγνώριση του προβλήματος και κάποια κίνηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Εγώ μπαίνω στη θέση των πατεράδων που λόγω της εθνικότητάς τους δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν πια τα παιδιά τους. Καταλαβαίνω ε, τον αγώνα σας και για μας πραγματικά έφτασε η ώρα ε, να αφήσουμε τα λόγια και να πιάσουμε τα έργα. Ωραία. Ο κύριος Βίντσε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικές αυτές οι ιστορίες που ακούσαμε από τους αναφέροντες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε να τις μοιραστείτε μαζί μας. Πολλά υπόθηκαν αλλά αυτό που μας εκπλήσει από άποψη Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι όχι μόνο το ότι δεν προβλέπεται κάποια λύση, αλλά και ότι προς ώρας δεν έχουμε καμία ουσιαστική απάντηση από την Ιαπωνική πλευρά. Εάν κατάλαβα καλά, ούτε γραπτή ούτε προφορική απάντηση έχει δοθεί ποτέ στα πλαίσια του ε, ε, διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ιαπωνίας. Ε, είναι δύσκολο να βρεθεί η λύση για την ώρα, γιατί δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτός ο διάλογος ο οποίος θα μπορούσε να μας προωθήσει, να προωθήσει τη σχέση αυτή. Ε, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, έκαναν ε, διαβήματα ε, Ιταλική κυβέρνηση κυρίως, ο, παρόλα αυτά πρέπει να υπογραφεί ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με μεταξύ των κρατών μελών που έχουν κοινό ενδιαφέρον και επομένως από κοινού να ασκήσουν πίεση προς την Ιαπωνική κυβέρνηση ως Επιτροπή Αναφορών ε, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βοηθήσουμε τους αναφέροντες. Καλωσορίζω, χαιρετίζω τα όσα είπε η Εύα στην παρέμβασή της. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε επιπλέον είναι να πούμε στην, ε, ε, στην αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ιαπωνίας ε, να ε, ε, γύρουν το ζήτημα αυτό εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επόμενη συνάντηση κορυφής. Προτείνω επίσης να κάνουμε μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Αυτό προτείνω στην Πρόεδρο. Είναι σημαντικό αυτό γιατί το θέμα είναι πολύ σημαντικό και πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε λύση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Κατανοώ βεβαίω στις πολιτιστικές διαφορές, αλλά παρόλα αυτά ζούμε σε ένα πολιτισμένο κόσμο ε, και η Ιαπωνία είναι από τις ηγέτιδες οικονομικές δυνάμεις. Ε, κατά την έννοια αυτή λοιπόν έχει και υποχρεώσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών. Άρα υποστηρίζω οποιαδήποτε ε, δράση ή πρωτοβουλία αναλυφθεί ε, και για μία ακόμα φορά εκφράζω τη συμπάθειά μου προς τους ε, αναφέροντες. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Μάεστρε Μαρτίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους αναφέροντες ότι τους υποστηρίζουμε πλήρως. Ε, ε, εμείς ε, πραγματικά μελετήσαμε πολύ προσεκτικά όλα αυτά που διαβάσαμε, που μας δώσατε, που μας είπατε το Κοινοβούλιο και αυτό πρέπει κάτι να κάνει. Δεν υπάρχουν εδώ ούτε δικαιολογίες, ούτε πολιτιστικά στοιχεία. κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση ε, δεν μπορεί η παράδοση ή η κουλτούρα να διευκολύνει ή να δικαιολογήσει παραβιάσεις δικαιωμάτων, κυρίως όταν αναφερόμαστε σε παραβίαση δικαιωμάτων ανηλίκων. Όπως είπαν και προλαλήσαντες συνάδελφοι, κυρίως ε, η κυρία Κόπακ ε, που υπέβαλε και προτάσεις, αλλά και αυτό που έλεγε και ο συνάδελφος Βίντσε και εγώ, θα ήθελα να προτείνω να κάνουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας γιατί εδώ έχουμε κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς επίσης και συγκεκριμένη βλάβη όσον αφορά ε, την ε, ε, σύμβαση δικαιωμάτων των παιδιών. Άρα, ε, από τη στιγμή που έχουμε και σχέσεις με την Ιαπωνία, εάν ε, κάνουμε μία έκθεση πρωτοβουλίας όπου θα αναφέρεται συγκεκριμένα αυτή η παραβίαση, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο. Γιατί είναι πολλές ε, οι οικογένειες, οι οποίες πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν παντρευτεί Ιάπωνες πολίτες και εμείς εδώ εδώ πραγματικά θα πρέπει να δεσμευτούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από το να πούμε ότι θέλουμε να σας στηρίξουμε. Βεβαίως να καταγγείλουμε την κατάσταση, αλλά να προτείνουμε και λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάιστρε. Επόμενος ομιλητής. Κυρία Σντάνοκα. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που αναδείξατε το θέμα αυτό ενώπιον μας. Εγώ δεν το γνώριζα. Δεν γνώριζα ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ελλειπής ενημέρωση του κοινού. Τα ζητήματα της αρπαγής ανηλίκων σε διάφορες περιστάσεις μας έχουν απασχολήσει σε πολλές περιπτώσεις εδώ στην Επιτροπή Αναφορών σε διασυνοριακές υποθέσεις αλλά επίσης και στο εσωτερικό των ε, κρατών μελών και τρίτων χωρών. Αλλά εγώ ως επιστήμονος, μαθηματικός είχα καλές σχέσεις με αυτή τη χώρα, με την Ιαπωνία, αλλά το πρόβλημα αυτό, αυτή την κατάσταση δεν την είχα ακούσει ποτέ. Επομένως, θα υποστηρίξω όλες τις προτάσεις που υπέβαλαν οι συνάδελφοί. Να αποστείλουμε επιστολή στην αντιπροσωπεία να φροντίσουμε τα στοιχεία αυτά να γίνουν γνωστά σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά επίσης θα έλεγα να κάνουμε και ε, επαφές με τον τύπο, δημοσιότητα. Και θα το ζητούσα και από εσάς, τους αναφέροντες, τους γονείς, να επιδιώξετε τη δημοσιότητα, να το μάθει ο κόσμος, γιατί νομίζω θα σας υποστηρίξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Εύη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να λάβω το λόγο για να υποστηρίξω αυτή την αναφορά, συμφωνώντας με πολλούς από τους συναδέλφους, όλους τους συναδέλφους. Κατά την παρουσίαση των υποθέσεων, των ιστοριών των προσωπικών από τους αναφέροντες, ε, αισθάνθηκα πολύ δύσκολα, πολύ, πολύ ε, μεγάλο βάρος, ε, ψυχολογικό, συναισθηματικό. Και θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τους αναφέροντες. Πιστεύω ότι είναι απολύτως απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση μετά από τόσες επιστολές, μετά από τόσες επικοινωνίες και διαβήματα, ουσιαστικά να μην έχει γίνει τίποτα. Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό και για να επαναλάβω αυτό που είπε και, ο κύριος, ε, και η κυρία Κόπατς. Θα πρέπει να συνεχίσουμε βεβαίως τις διπλωματικές επαφές, ε, τις επιστολές, να αναδεικνύεται το θέμα κάθε φορά από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κροατική Προεδρία θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις σχέσεις με την Ιαπωνία. Ε, θα ζητούσα όμως επίσης και η Επιτροπή μας να συντάξει μια επιστολή που να το ζητάει αυτό. Είναι γνωστό ότι εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εμπορικές συμφωνίες που έχουμε με τρίτες χώρες για να καταπολεμήσουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι είναι εδώ μια ευκαιρία να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι ενωμένη και με μια φωνή να προσπαθήσει να υπερασπιστεί αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όχι μόνο τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, αλλά και τα θεμελιώδη δικαιώματα των γονέων που παραβιάζονται διαρκώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Εύη. ο κύριος Άγος Σαλαμπά. Θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την αλληλεγγύη μου και την υποστήριξή μου προς τους αναφέροντες. Αυτές οι ιστορίες σοκάρουν και είναι πολύ δύσκολο όταν τις ακούει κανείς, αλλά θα πρέπει να επιθυμίσω ότι το 2016 η Επιτροπή Αναφορών είχε υιοθετήσει ψήφισμα, είχε προτείνει μάλλον ψήφισμα, για παρόμοιες καταστάσεις, παρόμοια προβλήματα που είχαμε εντοπίσει σε άλλες τρίτες χώρες, όχι μόνο την Ιαπωνία. Το Είχαμε αναδείξει ότι δεν γίνεται σεβαστός ο κανονισμός ε, Βρυξέλλες 2 θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα αυτών των γονέων. Ε, τα παιδιά τους μπορεί να μην ζουν πια στην Ευρώπη, αλλά παραμένουν Ευρωπαίοι πολίτες. Η ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών υποστηρίζει την αναφορά αυτή και ζητούμε μέσω του είπα του εκπροσώπου, του κ. Μπορέλ, να ασκήσουμε πίεση ακόμα μεγαλύτερη στην Ιαπωνία για όλες αυτές τις υποθέσεις για να δώσουμε μια λύση στα προβλήματα αυτών των γονέων από όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Άγγιο Σαλιμπά. Τελευταίος ομιλητής. Στα, στη μητρική μου γλώσσα. Πιστεύω ότι σεβόμαστε τις διαφορές. Μπορούμε να σεβαστούμε τις πολιτιστικές διαφορές των εταίρων μας, αλλά αυτό δεν μπορεί ποτέ να είναι μια δικαιολογία για να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και εν προκειμένου τα δικαιώματα των γονέων, πολιτών δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία και νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούμε στην Επιτροπή μας. Πιστεύω επίσης ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Πιστεύω πιο συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να ζητήσουμε ο κύριος Μπορέλ, ο υπότιτλος εκπρόσωπος, συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να στείλει επίσημη επιστολή στις αρχές της Ιαπωνίας δική του αρμοδιότητα είναι αυτές οι διεθνείς σχέσεις. Δεν αρκεί η πίεση που ασκεί μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, η πίεση πρέπει να ασκηθεί ακριβώς στο επίπεδο της ευρωπαϊκής διπλωματίας από την Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης. Οι αναφέροντες δύο λεπτά για τον καθένα. Ευχαριστούμε. Για να αποφύγουμε παραξηγήσεις διευκρινίζω πρώτον. Εδώ έχουμε μόνο ε, πατέρες εδώ, αλλά έχουμε και παραδείγματα μητέρων. Έχουμε μια Γαλλίδα μητέρα. Μέχρι ε, έχουμε και μια Αυστραλέζα που χωρίστηκε από τα παιδιά της. τα πολιτιστικά της Ιαπωνίας είναι προσχηματικά. Αν δούμε τη σύμβαση ε, για γενοκτονία ακόμα και τέτοιες περιπτώσεις καλύπτονται. Η ΠΟΗ επίσης αναγνώρισε την αποξένωση των παιδιών ως ε, πηγή προβλημάτων ψυχικής υγείας. Σε αυτή την περίπτωση, σε καθημερινή βάση υπάρχει αποξένωση. Ένα 155.000 παιδιά δεν έχουν σχέση με τους γονείς. Κάθε χρόνο αποξενώνονται στην Ιαπωνία. Τα τελευταία 20 χρόνια ε, ε, αυτό αθροίζεται σε 3 εκατομμύρια παιδιά. Γιατί οι περισσότερες αρχές δεν γνωρίζουν την κατάσταση. Διότι οι Ιάπωνες δικαστές ε, ε, χρησιμοποιούν συγκεκριμένη ρητορική για να δικαιολογήσουν και να νομιμοποιήσουν μια απαγωγή. Μπορείτε να διαβάσετε αποφάσεις των Ιαπωνικών ε, δικαστηρίων. Ποτέ δεν γίνεται λόγος για απαγωγή εκεί. Δέχονται την κατάσταση αλλά δεν την καταδικάζουν. Μια σύντομη προσθήκη. Η δική μου περίπτωση είναι η σαφέστερη από τότε που επικύρωσε τη συμφωνία η Ιαπωνία. Έχω, μοναδική, έχω μόνο εγώ την επιμέλεια, ε, έχω μέτρα επιβολής ε, υπέρ μου, αλλά τι άλλο να ζητήσει κανείς ε, επισήμως, τα έχω όλα. Αλλά ακόμα τα παιδιά μου δεν έχουν επαναπατριστεί. Πώς είναι δυνατόν ε, να φέρετε έτσι μια χώρα που δηλώνει δημοκρατική. Μπορεί να μην ξαναδώ τα παιδιά μου τα επόμενα 15-20 χρόνια. Κάθε φορά που θα βλέπουν αυτό το βίντεο θα είναι ευγνώμων ε, προς εσάς. Εξ ονόματος των παιδιών μου και εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πρέπει να δράσουμε άμεσα. Τα παιδιά μου είναι θύματα εγκληματικής ενέργειας. έχουν κακοποιηθεί. Δεν μπορούμε να περιμένουμε την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής πρέπει να ληφθούν μέτρα χθες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε μία μέρα ακόμα. Διαφωνώ με κάτι που άκουσα σήμερα ότι είναι, υπάρχουν διαφορές κουλτούρας. Αν υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές, γιατί πας και κυρώνεις διεθνή συμφωνία. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών κυρώθηκε από την Ιαπωνία. Δέκα χρόνια τους πήρε αν δεν συνάδει η σύμβαση αυτή με τους εθνικούς κανόνες, μην πας να κυρώσεις και να υποκρίνεσαι ότι σέβεσαι τα δικαιώματα των παιδιών. Υποχρεούται η Ιαπωνία να συμμορφωθεί ένα άλλο θέμα. Αν η Ιαπωνία δεν μπορεί να σέβεται τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών όπως ορίζονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τι πιστεύει το Κοινοβούλιο, θα σεβαστεί τη Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας την επόμενη φορά που θα μας χτυπήσει η κρίση, αν δεν μπορεί να δεχτείς τα δικαιώματα των παιδιών, πώς θα δεχτείς εμπορικές συμφωνίες όταν δεν έχεις την πολυτέλεια να το κάνεις. Εγώ θα ανησυχούσα πολύ ως ο Ευρωπαίος νομοθέτης σχετικά με την ικανότητα και δυνατότητα της Ιαπωνίας να σεβαστεί οποιασδήποτε συμφωνίες. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ε, δράσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα. Και μην εμπιστεύεστε στους Ιάπωνες όταν λένε ότι το εξετάζουν το θέμα. Το εξετάζουν εδώ και 20 χρόνια. Χρειάζονται να τους ε, ε, δώσουμε κανένα λάκτισμα. Ε, δεν, μπορούμε, δεν έχουμε εναλλακτικέ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχουμε γονεϊκά δικαιώματα, αλλά όταν πάμε να επισκεφθούμε τα παιδιά μας αύριο, αύριο θα έρθει η αστυνομία και θα μα βάλει φυλακή, Όπω έγινε σε, έναν Αυστραλό που πήγε στην Ιαπωνία 45 μέρε, ε, και ήταν σε κοινό χώρο, σε ένα χώρο κατοικιών, ε, συνελήφθη. Ε, πάμε να δούμε τα παιδιά μας, δεν τα βλέπουμε και μας απειλούν με φυλάκιση, ε, τιμωρία. Ε, κάνουν προσφυγές στα δικαστήρια. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Αν μπορείτε να κάνετε κάτι, κάντε το γρήγορα, γιατί τα παιδιά μας μεγαλώνουν και σε λίγο θα ξεχάσουν ποιοι είναι οι Ευρωπαίοι γονείς τους. Σας ευχαριστώ. Είμαστε πολύ απελπισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ τρομερά όλα αυτά. Τώρα, προτείνω πολύ συγκεκριμένα βήματα. Πρώτον, πρέπει να ανοίξουμε τη διαδικασία. Δεύτερον, πρέπει να απευθύνουμε επιστολή στον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης και να ζητήσουμε συγκεκριμένες δράσεις. Τρίτον, μπορούμε να απευθύνουμε επιστολή στην Ιαπωνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ιάπωνα Πρέσβη και τέλος προτείνω να εγκρίνουμε ένα σύντομο ψήφισμα επί του θέματος. Συμφωνείτε? Εμείς συμφωνούμε απόλυτα. Και το ΕΛΚ στηρίζει απόλυτα τις προτάσεις και στην Ολομέλεια την ε, και θα, θα, ε, ζητηθεί να συζητηθεί από την Ολομέλεια το θέμα και θα ενημερώσουμε και την κοινοβουλευτική μας ομάδα εδώ για το ζήτημα. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Παρακαλώ, Ινάσιο. Συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους. Δεν μπορούμε όμως να περιμένουμε μέχρι να αντιδράσει η αντιπροσωπεία. Πρέπει παράλληλα να ζητήσουμε από τον πρόεδρο όλοι να αναλάβει δράση γρήγορα με την Κομισιόν διότι αν υπάρξει ε, θέμα κυρώσεων ε, σε σχέση με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, τότε θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Μην περιμένουμε μέχρι την επόμενη Ολομέλεια να μπει το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Μπορούμε μέσω Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιταχύνουμε τη διαδικασία, να ευαισθητοποιηθεί και η Κομισιόν και να ληφθούν μέτρα νωρίτερα. χωρίς να αποκλείουμε τα άλλα που είπατε. Ωραία. Θα ενημερώσουμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά και θα ε, συζητήσουμε και στην επόμενη Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε την συνεδρίαση στο σημείο αυτό. Καλή σας όρεξη.